So good afternoon. I'm speaking now in German. Σας απόγευμα και θα συνεχίσω γερμανικά. Φορέστε τα ακουστικά σας. Παρακαλώ. Uh, Έχουμε χάσει απολέσει ένα συνάδελφο που επέστρεψε στην εθνική πολιτική. Ο συνάδελφος Σόινια αποχώρησε από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι τώρα μέλος στο Φινλανδικό Κοινοβούλιο. Και ελπίζω στο πλαίσιο της εθνικής εργασίας του βουλευτή ως βουλευτής να μην ξεχάσει τις ευρωπαϊκές ιδέες και τα ιδανικά και να αναζωογονηθούν αυτά εκεί. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το νέο του αξίωμα που είναι και σημαντικό και για τη Φινλανδία. Έχουμε την κατάσταση που μπορούμε να χαιρετήσουμε έναν νέο συνάδελφο από αυτή τη χώρα, τον συνάδελφο Σαμποφέρο. Καλώς ήρθατε. Θα είσαστε ένας καλός συνάδελφος ελπίζω. Και εκείνος είναι στην ομάδα των ε, SD. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διευρύνουμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα με την εκλογή, την εκλογή του νέου αντιπροέδρου. Επειδή ο κύριος Σόνι αποχώρησε ακριβώς. Μπορούμε να διευρύνουμε την ημερήσια διάταξη με αυτό το σημείο, παρακαλώ. Όλοι πήρατε αυτή την ειδοποίηση έγκαιρα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτής της εκλογής για απόψε. Μαρία παρακαλώ, η Μαρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Προσέξτε, εγώ δεν πήρα καμιά πληροφόρηση ότι σήμερα θα έπρεπε λέει να ψηφίσουμε για αυτή την αλλαγή, για αυτό το αξίωμα. Θα ζητούσα αν είναι δυνατόν να το αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής. Ε, δεν ειδοποιηθήκατε, λέτε ότι θα ψηφίζαμε σήμερα, όμως πήρατε την ειδοποίηση ότι η ομάδα αυτή για τον αποχωρήσαντα Σόνι προτείνει τον κύριο Πρέρο και είναι η πρώτη συνεδρίασή μας απόψε και νομίζω απόψε μπορούμε να το διευθετήσουμε. Δεν χρειάζεται να το αναβάλουμε. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Αν μπορεί να μου αναφέρει ένα λόγο, γιατί να συμβεί αυτό, γιατί να γίνει αυτό, παρακαλώ να μου το εξηγήσει. Ο κύριο Τάκουλα έχει τον λόγο πρώτο. Παρακαλώ, κύριε Τάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να από πλευρά μου να πω πρώτα απ' όλα ότι καλωσορίζω τον καινούριο συνάδελφο, τον καλωσορίζω θερμά. Πρόκειται με τη διαδικασία εκπροσώπησης DOND, με την αρχή DOND. Με αυτή την αρχή θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Θέλουμε να τηρείται αυτή η αρχή από το Ευρωκοινοβούλιο. Στη Μαρία μπορώ να πω ότι τον κύριο Πέρο τον γνωρίζω καλά. Είναι ένα πραγματικά αξιόλογος συνάδελφος και επικοδομητικός όσον αφορά το πνεύμα συνεργασίας. Ως αντιπρόεδρος μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά και το χαιρετίζω αυτό να γίνει. Να το κάνουμε έτσι λοιπόν παρακαλώ. μικρόφωνο. Θα ήθελα να υποστηρίξω ε, τη Μαρία γιατί ούτε εγώ έλαβα ειδοποίηση. Αν μπορούσαμε να το αναβάλουμε μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, τουλάχιστον μέχρι αύριο, για να έχουν τη ε, δυνατότητα οι αντιπροσωπείες να το εξετάσουν. Θα μπορούσα να αφήσω να ψηφίσουμε απόψε. Θα είχαν οι υπέρ πλειοψηφία. Αλλά είμαι ευγενή. Αν χρειάζονται μία μέρα παραπάνω οι συνάδελφοι οι σοσιαλιστέ, να το κάνουμε έστω και αυτή τη φορά με την αρχή των. με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το αναβάλουμε λοιπόν για αύριο. Για αύριο είμαι πρόθυμη να μην συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα. Να, για το αναβάλουμε όμως επαόριστον δεν το δέχομαι. Το δέχομαι μόνο μέχρι αύριο. Παρακαλώ. Μαρία. Bueno. Λοιπόν, δεν μου φάνηκε ότι ζητούσαμε κάτι το αξιοπερίεργο. Είχαμε μια ημερήσια διάταξη που είχε προταθεί. Υποβάλλεται μια πρόταση αλλαγή τη ημερήσια διάταξη. Πρόκειται την εκλογή νέου αντιπροέδρου. Και γνωρίζοντα ε, αυτά τα οποία ζητήσαμε, το μόνο που ζητήσαμε κάποιε ώρε να έχουμε στη διάθεσή μα, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ένα μεταξύ μα. Ξέρετε απόλυτα πρόεδρε, τέλεια εκείνο που είχαμε ψηφίσει στο παρελθόν. Ξέρετε τι εκστρατεία έκανε το κόμμα αυτό στη Φινλανδία, ξέρετε για τις αρχές που προάσπισε, που δεν είναι ακριβώς οι δικές μας αρχές. Και το μόνο που θέλουμε είναι να συζητήσουμε κάπως αυτό το θέμα. Καλό λοιπόν είναι και σας ευχαριστώ γι' αυτό να το αναβάλουμε για αύριο, να ρυθμιστεί αύριο αυτό. Ευχαριστώ. Δεν έχει τον λόγο. Σε συμπαθώ, αλλά δεν είναι. Δεν σου έχω δώσει τον λόγο. Εγώ θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσει κανεί περαιτέρω. Δεν είναι συζήτηση αυτή που ξεκινήσαμε. Εντάξει, το δέχτηκα ότι επιθυμείτε να ψηφίσουμε αύριο. Τελεία και παύλα. Όταν είπατε όταν είχατε την παρέμβασή σα την πρώτη είπατε την επόμενη μα συνεδρίαση. Ε, λοιπόν, όχι την άλλη επόμενη συνεδρίαση άλλοτε, αλλά αύριο. Θα έχετε χρόνο και θα μπορούμε μέχρι αύριο να ψηφίσουμε. Δεν χρειάζεται τώρα να αρχίσουμε και να τραβάμε διαχωριστικές γραμμές και να διαχωριζόμαστε. Είμαστε πρόθυμοι, αύριο θα γίνει αυτό, έχετε χρόνο να προβληματιστείτε, αύριο το πρωί σε 9 θα το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ για την κατανόηση Ευχαριστώ και για την κατανόηση σε σχέση με τον νέο συνάδελφο. Έχουμε κανονισμούς, πρέπει να τους στηρίσουμε όταν πρόκειται για αλλαγή. Πρέπει να προσπαθήσουμε χωρίς γραφειοκρατική επιβάρυνση να τα ρυθμίζουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Έγκριση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης. Αν έχετε κάποιες αντιρρήσεις ή ενστάσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας να μας, να μας γνωστοποιήσετε τις αντιρρήσεις σας. Αλλιώς τα πρακτικά θα θεωρεί ότι κυρώνονται. Περνάμε στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης. Υπενθυμίζω ότι βρίσκεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Κάθε ένας μπορεί να την παρακολουθήσει και μέχρι την Φινλανδία. Ελπίζουμε ότι ο συνάδελφος Σόνι παρακολουθεί. Αν παρακολουθεί του ευχόμαστε καλύτερη συνειδητοποίηση ευρωπαϊκών θεμάτων από ό,τι κατέδειξε σε σχέση με τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Όλοι θα θέλαμε να βοηθήσουμε. Και ίσως και ο νέος συνάδελφος που εδώ παρίσταται μπορεί κάπως ε, να διαβιβάζει τα θέματα αυτά προς τον συνάδελφο Σόνι στην Φινλανδία που τον εκτιμούμε όλοι και που πραγματικά με, ιδιαίτερη, με ιδιαίτερα εύγλωτο τρόπο θα μπορούσε αυτό να ε, γίνει με αυτόν τον τρόπο δεν ξέρω γιατί χρειάστηκε αυτή η διαδικασία. Έχουμε ε, διερμηνία, έχουμε όλες τις γλώσσες. Εκτός, εκτός διορθώνω λέει η Πρόεδρος, τσεχικά, λετονικά, λιθουανικά και ε, μαλτέζικα. Όλα τα άλλα είναι διαθέσιμα στις ε, μεταφράσεις. Σύντομα θα ήθελα να σας επεξηγήσω τι κάναμε τον τελευταίο, το τελευταίο διάστημα, τι έγινε. Είχαμε την ετικέτα Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς, αυτή την ονομασία. Βρίσκεται καθοδόν σε σωστή πορεία. Η κυρία Παγιατέλη, η, η συγγήτρια και εγώ είχαμε εντολή να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε πώς το λέμε σε μια πρώιμη συμφωνία πρώτης ανάγνωσης, έγκαιρα στην πρώτη ανάγνωση. Το προσπαθήσαμε, το καταφέραμε και τώρα καταφέραμε να διευθετήσουμε αυτό το θέμα. Όλοι οι σκιώδεις εισηγητές ενεπλάκησαν, πάντα ενημερωνόντουσαν, κανείς δεν μπορεί να πει ότι κάναμε κάτι χωρίς να εμπλέκονται εκείνοι. Την τελευταία εβδομάδα το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας ε, και Πολιτισμού κατέληξαν σε μια πολιτική συμφωνία για αυτό το συμβαστικό κείμενο μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και το Συμβούλιο τώρα θέλει επίσημα πλέον να εκφράσει την άποψή του τον Ιούλιο. Με επίσημο τρόπο θα ψηφίσουν και θα εγκρίνουν. Και όταν θα έχει ψηφιστεί και διευθετηθεί τον Ιούλιο, τότε το Σεπτέμβριο από εμάς στην πρώτη ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα τεθεί προς ψηφοφορία προσέγγιση. Διευθετήθηκε αυτό να έχετε εμπιστοσύνη ότι η ιδέα αυτή της ονομασίας ευρωπαϊκής κληρονομιάς προχώρησε και ότι πραγματικά έτσι θα φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη ένα βήμα και στην Φινλανδία ελπίζω με την ετικέτα, με την ονομασία Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς και στη Φινλανδία ελπίζουμε ότι θα έχουμε επιτυχία. Μια αντιπροσωπεία επιπλέον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Τούρκου και στο, στο Ταλίν θα θέλαμε τους συναδέλφους, τους συναδέλφους να δώσουμε την ευκαιρία να πούν δύο λόγια για αυτή την αποστολή. Αυτή τη στιγμή ο συνάδελφος είναι απασχολημένος, θα ήθελε να παρέμβει. Παρακαλώ, έχεις τον λόγο συνάδελφε. Ξέρεις για ποιο θέμα, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μπορούμε να πούμε ότι είχαμε μια πολύ επιτυχή και επικοδομητική εβδομάδα στο Τούρκου και στο Ταλίν. ήταν ε, ιδιαίτερα βαρύ το πρόγραμμα και στις δύο αυτές περιοχές ε, με πολλές δραστηριότητες. Ε, όλοι οι συμμετέχοντες επέδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Εγώ προσωπικά αλλά και στους συνάδελφους που μίλησα είπαμε ότι Θέλαμε πραγματικά να πάμε εκεί. Ξέρουμε ότι ο συνάδελφος ο Χάνου είναι από το Τούρκου και μας είχε προετοιμάσει ένα πολύ ευχάριστο βράδυ. Καταφέραμε να, ακόμα και να είχαμε τη δυνατότητα να τραγουδήσουμε ακόμα και φιλανδικά ε, παραδοσιακά τραγούδια. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που χαρακτήρισε το Τούρκο ήταν ότι είχε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα και καταφέραμε να δούμε πολλά από τα όσα εξελίσσονται αυτή τη στιγμή εκεί. Αν το συγκρίνουμε με το Ταλίν, μπορούμε να πούμε ότι εκεί υπήρχε πολύ περιορισμένος ο Παρ' όλα αυτά κατάφεραν να βρουν να καταλήξουν και να διοργανώσουν ιδιαίτερα ε, δημιουργικές εκδηλώσεις. Δηλαδή δεν γυρνούν τα πάντα γύρω από το χρήμα αν και είναι πολύ σημαντικό, το ξέρω. Αλλά όταν ε, δημιουργείς έμπνευση, ε, τότε μπορείς να καταλήξεις σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία εκεί. Ε, συζητήσαμε και με τις οργανώσεις εκεί για την εμπειρία τους μέχρι τώρα και τι μπορούν να κάνουν μέχρι την επόμενη φορά ε, και πώς να στηρίξουν ε, τους επόμενους υποψηφίους. Γενικότερα όμως ήταν πολύ επικοδηματική εμπειρία. Μαρία. Μαρία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να προσθέσω και εγώ επίσης τα λόγια του συναδέλφου ότι είμαστε μέρο αυτής της αντιπροσωπείας για το, την αποστολή αυτή που ήταν πολύ επιτυχής και στέφηκε με επιτυχία. Να συγχαρώ τον Άννο, διότι παρότι μπορεί να έχουμε διαφορές σε κάποια θέματα, η διοργάνωση στο Τούρκου ήταν εξαιρετική η πρόσκληση, η δική του προσωπική πρόσκληση επίσης και ευχαριστώ πολύ για αυτή. Και θέλω να ευχαριστήσω και το Τούρκου και το Ταλίν ως πόλεις για ένα πράγμα ιδιαίτερα, διότι αυτές οι δύο πόλεις ενέπλαξαν, ενέπλεξαν πάρα πολύ τους πολίτες τους σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θεμελιώδης αξία αυτή. Και θέλω να συγχαρώ για το έργο που έγινε. Να ευχαριστήσω όλους που κατέστησαν ε, δυνατό να γίνει αυτή η αποστολή. Ευχαριστώ. Είναι τόκο. Σύντομα παρακαλώ, εσείς. Σε ευχαριστώ. Είχα πάει στο Τούρκο, αλλά πιο πριν ε, είχα ε, ένα πράγμα διασφαλίσει σε σχέση με το Τούρκο, ένα σημαντικό πράγμα που δείχνει ότι δεν χρειάζεται πάντα να είναι μια μεγάλη πόλη εκείνη που θα έχει τεράστιες υποδομές ώστε να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το υπόδειγμα, το πρότυπο του Τούρκου κατέδειξε εδώ ότι είναι ενδιαφέρουσα η δυνατότητα να υπάρχουν πολιτισμικές, πολιτιστικές δυνατότητες σε μιας μικρότερης πόλης και ένας αντίστοιχος προϋπολογισμός με κονδύλια, ώστε δεν χρειάζεται να είναι μητρόπολη η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Νομίζω μπορούμε να πούμε αυτό ότι το δίκτυο των ευρωπαϊκών πρωτεύουσών στο μέλλον θα πρέπει να υποστηριχθεί, γιατί έχουμε μεγάλο δυναμικό και έρχονται πολύ καλά σε επαφή και συνεργάζονται μαζί τους. Κύριε, μεγάλη αξία για το μέλλον αυτό να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. πρόεδρο, ευχαριστώ. Θέλω να υπενθυμίσω στην τελευταία συνεδρίαση στο Στρασβούργο το θέμα του Σαράγεβου. Επιτυχώς το ολοκληρώσαμε. Είχαμε ομόφωνα, δεν ξέρω αν όχι ομόφωνα, τουλάχιστον με συντριπτική πλειοψηφία είχαμε ψηφίσει για το 2014 ως εξαίρεση μια τρίτη πολιτιστική πρωτεύουσα να κατονομαστεί το Σαράγεβο με την επέτειο από το 1914-2014 από την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τότε, τον 20ο αιώνα. Και η χαρά που δημιουργεί αυτή η απάσταση είναι μεγάλη. Όμως πρέπει τώρα να πείσουμε το Συμβούλιο ότι αυτή την εξαίρεση πρέπει να την εγκρίνει το ίδιο το Συμβούλιο. Δώσαμε την υπόσχεσή μας, τον λόγο μας, ότι την απόφαση εκείνη που πήραμε για το 2014, για το 2017 θα έχει συνέπειες. Παρακαλώ στους συναδέφους, στους συναδέλφους, τους υπουργούς τους ε, να ασκήσουν πίεση, να είναι υπέρ αυτής της εξαίρεσης. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν όλα αυτά τον Ιούνιο ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε έγκαιρα. Παρακαλώ να μην βασιζόμαστε ότι έγινε αυτό με αυτόν τον τρόπο και έτσι θα περάσει και θα εγκριθεί, να ασκήσουν όλη την επιρροή και την πίεσή τους. Ε, το ζητώ αυτό για να το πετύχουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Περνάμε στο σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Το σύστημα ευρωπαϊκών σχολείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε όλοι, τα ευρωπαϊκά σχολεία ιδρύθηκαν ώστε τα παιδιά των υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων στη μητρική τους γλώσσα να μπορούν να εκπαιδεύονται και εντωμεταξύ έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και είναι ανοιχτά τα σχολεία και για άλλου, εκτό δηλαδή των παιδιών των υπαλλήλων. Υπάρχουν προβλήματα πάσης φύσεως και του διορισμού των ε, δασκάλων και καθηγητών, χρηματοοικονομικά προβλήματα. Έχουμε παρακαλέσει τον συνάδελφο Καβαντά, τον εισηγητή μα, να ασχοληθεί με το θέμα και να συντάξει μια έκθεση. Αν δεν απατώμε, υπήρξε συζήτηση σήμερα το πρωί με εκπροσώπου, με τον Γενικό Γραμματέα ε, των Ευρωπαϊκών Σχολείων, με τον Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω υπήρχε και η δυνατότητα να ε, παρακολουθηθεί αυτή. Δίνω τον λόγο στον συνάδελφο Καβαντά να μας εκθέσει για την έκθεσή του τα σχετικά. Έχετε τον λόγο κύριε Καβαντά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εξαιρετική του συνεργασία το σύνολο των συναδέλφων της Επιτροπής μας. Η παρασκευαστική δουλειά ήταν ε, τελικά κακοφόρα στα πλαίσια της τελευταίας συνάντησης των σκιωδών εισηγητών. Δεν υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία ανατίθενται, αλλά δεν πρέπει να είναι κανείς πολύ αισιόδοξο. Θα δούμε σε ποιο βαθμό οι τροπολογίες τις οποίες αναμένουμε θα κατατεθούν. Πρόκειται για ένα συνθετικό κείμενο, δεν είχα την επιλογή, θα σας εξηγήσω γιατί. Περιοριστήκαμε σε 6.000 γράμματα, χωρίς χώρους μεταξύ τους για τεχνικούς λόγους. Είχαμε δύο επιλογές, ή να καταργήσουμε κάποιες παραγράφους και να αφήσουμε έξω σημαντικά κομμάτια, ή να διατηρήσουμε με συνθετικό τρόπο κάποια σημεία τα οποία θα ήθελα να συγκρατήσουμε ε, μένοντας πάντα πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Γι' αυτό έχετε λοιπόν μια τέτοια συνθετική έκθεση μαζί σας. Οι τροπολογίες έτσι και αλλιώ θα μας επιτρέψουν να μεγαλώσουμε, να μεγενθύνουμε την εργασία αυτή. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών μέσα Ιουνίου, ψήφος στην Επιτροπή μας 14 Ιουλίου και μπορούμε το Σεπτάμβριο στη δεύτερη Ολομέλεια να είμαστε έτοιμοι. Τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν αποδείξει την παιδαγωγική τους χρησιμότητα σε επίπεδο διαπολιτισμικότητας και εκμάθησης γλωσσών. Θα μπορούσαν λοιπόν να χρησιμεύσουν σαν πρότυπο και για τα εθνικά επίπεδα. Αναφέρομαι στην έκθεση στην οργάνωση του ίδιου του συστήματος, της προώθησης του Ευρωπαϊκού Μπακαλωρεά, της αναδιάρθρωσης των δημοσιονομικών προβλημάτων, της αυτονόμησης ε, των ίδρυμάτων και των παιδαγωγικών ρυθμίσεων που θα είναι απαραίτητες για την προσαρμογή του συστήματος και για την ε, δημιουργία ενός πιστοποιητικού τέλους σπουδών εκτός από τον μπακαλωρεά για παιδιά τα οποία θα πρέπει να φύγουν νωρίτερα. Ταυτόχρονα υποστηρίξαμε στην Ζουριντικ τον αντιπρόσωπό μας για να υπάρξει σωστή νομική βάση για τη λειτουργία των σχολείων έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμεύσει και για άλλους μαθητές, όχι μόνο αυτούς που εργάζονται στα ευρωπαϊκά όργανα. Επιμένουμε λοιπόν στην οργάνωση και την ανάπτυξη του συστήματος των σχολείων αυτών και την ανάγκη να προωθήσουμε το Ευρωπαϊκό Μπακαλωρεά που έχει εξαιρετική φήμη και να αυτονομήσουμε τα Ιδρύματα. Θα ήθελα να θέσω κάποια σημεία τα οποία από ό,τι φαίνεται παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς, τα ευρωπαϊκά σχολεία δημιουργήθηκαν το 1953. Είναι κάτι το καινοτόμο, που γεννήθηκε από την ανάγκη να πάνε σχολείο τα παιδιά τα οποία είχαν έρθει να εργαστούν εδώ στη μητρική τους γλώσσα, οι γονείς τους είχαν έρθει εδώ στη μητρική τους γλώσσα. Επιβάλλονται κάποιες βασικές αρχές. Καταρχάς διδασκαλία στη μητρική γλώσσα. Δεύτερον, μια πολύγλωση εκπαίδευση. Τρίτον, διδασκαλία γλωσσών που δίδεται από καθηγητές, χορηγείται από καθηγητές που προέρχεται από τα εθνικά συστήματα εκπαίδευση. Τέταρτον, δυνατότητα σύνθεσης ενός προσωπικής φύσεως σχολικού προγράμματος. Πέμπτον, ευνόηση της πολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας, κάτι το οποίο είναι η βάση για ε, μια πολιτιστική ευρωπαϊκή πατρίδα. Ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων δεν είναι πλέον αυτός που θα έπρεπε για μια Ευρώπη των 27 διαπιστώνουμε ότι η χρηματοδότηση βασίζεται στη συνεισφορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πόρων τα οποία, οι οποίοι συλλέγονται από τα, χρήματα που κατατίθεται για την εγγραφή των φοιτητών. Θα πρέπει εδώ να το δούμε διαφορετικά το πρόβλημα. Υπάρχει ένα θέμα σχετικό με την απόσπαση των καθηγητών. Κάποια κράτη-μέλη δεν βλέπουν να είναι αντίστοιχο ο αριθμός των καθηγητών που αποσπώνται με τον αριθμό των φοιτητών. Από το 2004, αναγλωσσικό τμήμα, ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται και πολλοί ε, μαθητές αναγκάζονται να πηγαίνουν σε άλλα σχολικά τμήματα, γλωσσικά τμήματα, κάτι το οποίο απαιτεί πρόσληψη περισσότερων καθηγητών. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη που δεν δίδουν καθηγητές να συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό του σχολείου. Θα πρέπει επίσης για να σεβαστούμε τη φιλοσοφία λειτουργία και το δικαίωμα των παιδιών να παίρνουν τη διδασκαλία που δικαιούνται στη γλώσσα τους, θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα σχολικά γλωσσικά τμήματα εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών, ο ικανός αριθμός μαθητών. Υπάρχει θέμα κατανομής των μαθητών αυτών και αυτό και η οικονομική κρίση δεν θα πρέπει να φύγει ε, τους μαθητές, ιδιαίτερα τους μαθητές οι οποίοι έχουν προβλήματα. Λοιπόν, αυτά τα θέματα έχουν και πολιτικό βάρος και τεχνικό βάρος. Είναι βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διατύπωση των τροπολογιών. Συνάδελφοι, δεν έχω κάτι άλλο, είμαι στη διάθεσή σας, θα σας ακούσω και θα συζητήσω γιατί όχι. Σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Νοφεγγάης παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία χρειάζονται κάποια μεταρρύθμιση και νομίζω όλοι συμφωνούν επ' αυτού. Πιστεύω επιπλέον και όταν ζήτησα να παρέμβω σε σχέση με αυτή την έκθεση πιστεύω και πρέπει να το πω αυτό ότι γίνεται για τον εξή λόγο επειδή πιστεύω ότι τώρα πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το έργο που επομιζόμαστε σε αυτή τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας για την έναρξη κάποιων μεταρρυθμίσεων να μην κάνουμε κάτι το οποίο τις βασικές αρχές θα τις παραβίαζε ή τις ιδρυτικές αρχές αυτών των σχολείων θα τις παραβίαζαν. Είναι σαφές ότι υπάρχουν μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα, εποχή λιτότητας, πρέπει να γίνουν εξοικονομήσεις ε, χρημάτων. Αν τώρα εδώ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση ε, προς μια κατεύθυνση εξετάσουμε τις τροπολογίες Συνιστώ του συναδέλφους η αφετηρία μας να είναι οι μικρότερες εντός εισαγωγικών γλώσσες με τον έναν ή άλλο τρόπο να διασφαλιστούν ως γλώσσες διδασκαλίας. Διότι για μένα είναι μια βασική αρχή αυτή της ιδρυτικής σκέψης, ίδρυσης ακριβώς και συγκρότησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Απευθύνω έκκληση όταν εδώ εργαζόμαστε επ' αυτού να ληφθεί υπόψη και να υπάρξει κατανόηση που θα δείξουμε για αυτό το θέμα αυτής της αρχής το Κάποιες ώρες μόνο γίνονται γλωσσικών μαθημάτων σε κάποιες γλώσσες. Όμως Παρ' όλα αυτά είναι γλώσσες αυτές που διακυβεύονται και αντιμετωπίζουν κίνδυνο που ελοχεύει να εξαφανιστούν από το πρόγραμμα. Να μην το κάνουμε λοιπόν αυτό, να μην αφήσουμε να γίνει, να υπερασπιστούμε αυτές τις γλώσσες. Ε, ξέρουμε όλοι τι σημαίνουν οι γλώσσες για μας. Ξέρουμε και τι σημαίνει η γλώσσα μας για την πατρίδα μας και τι σημαίνει αυτό πολιτισμικά για τον, την εκλογική μας περιφέρεια, για μας τους ίδιους. Θα συνιστούσα λοιπόν να πετύχουμε ομοφωνία και συνένεση για αυτές ε, τις ώστε να διασφαλιστούν τα κονδύλια ώστε αυτές οι γλώσσες να διασφαλιστούν. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα κατά πρώτον να ευχαριστήσω τον ίδιο τον κύριο Καβαντά για μια πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για την διοργάνωση του, της σημερινής Τράπεζα ήταν μια σημαντική συνεισφορά, διότι πολλοί συνήθαν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί που καθημερινά ασχολούνται και έχουν επάγγελμα αυτό το θέμα της διδασκαλίας στα ευρωπαϊκά σχολεία. Είτε ήταν δάσκαλοι, είτε πρόσωποι γονέων, είτε από τη διεύθυνση. Η συζήτηση ήταν πολύ επικοδομητική. Κάποιε διαφορετικέ απόψει επί διαφορετικών θεμάτων αναφέρθηκαν. Θα ήθελα να αναφέρω ότι χρειάζονται, λέει, περισσότερα κονδύλια. Αυτό το λέει και η δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όλο και περισσότερα κονδύλια θα χρειαζόμαστε χρηματοοικονομικά. Διότι όταν και αν θα έχουμε περισσότερα κονδύλια θα μπορούμε περισσότερα πράγματα να κάνουμε. Αυτό ισχύει φυσικά και για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Υποστηρίζω την άποψη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη πειθαρχία από τα κράτη-μέλη ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους με τον δέοντα τρόπο. Πρόκειται για τους ίδιους τους πολίτες εκείνων των χωρών που πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και να καλλιεργούν τη γλώσσα τους εναντί των πολιτών τους που προσέρχονται στα ευρωπαϊκά σχολεία. Η κυβερνήσεις και οι χώρες πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνες τους και να ανταποκριθούν να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Σημαντικό είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας στις γλώσσες εκείνες που τις αποκαλούμε μικρότερες γλώσσες. Όχι μόνο αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά, αλλά και τις άλλες γλώσσες οπωσδήποτε. Όταν χρησιμοποιείται το επιχείρημα ότι υπάρχουν λίγα λέει παιδιά σε αυτά τα σχολεία, αυτό το επιχείρημα δεν ευσταθεί δεν είναι βάσιμο. Διότι πολύ συχνά συμβαίνει αυτό να χρησιμοποιείται προσχηματικά ως επιχείρημα επειδή για αρκετές γλώσσες λέει δεν υπάρχουν αρκετοί μαθητές και έτσι λοιπόν δεν θα διδάσκονται αυτές οι γλώσσες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο σημαντικό να μιλάνε όλοι αγγλικά, αλλά είναι και σημαντικό στι υπόλοιπε άλλε γλώσσε να υπάρχει δυνατότητα διδασκαλία. Ιδιαίτερα όταν έχουμε γλώσσε ε, μεταναστών που θέλουμε να υποστηρίξουμε τη διδασκαλία του, αυτέ οι μικρότερε γλώσσε δεν πρέπει να αγνοούνται, δεν πρέπει να αμελούνται με κανένα τρόπο. Επιπλέον θα πρέπει να ανοιχθούμε και εναντίον άλλων θεσμικών οργάνων όσον αφορά την ίδια την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να ανοιχθεί σε σχέση με αυτό. Έχουμε προβλήματα με τη χρηματοδότηση. Όταν εμείς για παράδειγμα με το ΝΑΤΟ ερχόμαστε σε επαφή και συνεννοούμαστε ή με άλλα θεσμικά όργανα, αυτά τα θεσμικά όργανα έχουν και εκείνα εκπροσώπηση ή θηγατρικά γραφεία σε πόλεις όπου χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζονται υποστήριξη. Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω την ιδέα της αναγνώρισης, της αναγνώρισης του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου Λυκείου είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην περνάνε, να μην αναγκάζονται να υποστούν πρόσθετες εξετάσεις επιπλέον από πλευράς αρχών κρατών μελών. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να συζητήσουμε. Αυτά όμως είναι αυτά τα οποία θα ήθελα να πω και πακούμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Η κυρία Παλιατέλη παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα, παίρνω περισσότερο το λόγο για να συγχαρώ τον κύριο Καβαδά ε, για την εξαιρετικά εμπεριστατωμένη ε, έκθεση ε, στην οποία ομολογώ ότι δεν ξέρω αν θα βρίσκα τρόπους να κάνω τροπολογίες. αν υπάρχουν σημεία να δεχτούν τροπολογίες. Θέλω μία ερώτηση η οποία έχει σχέση με την ουσία. Το Ανώτατο Συμβούλιο ενέκρινε το Μάιο του 2009 ανάμεσα στις άλλες προτάσεις και το άνοιγμα του συστήματος σε σχολείου τύπου 2 και 3 ε, αυτό γίνεται με ποια διαδικασία. Εθνικά σχολεία τα οποία προσαρμόζονται στο ευρωπαϊκό σύστημα, ε, στο σύστημα των σπουδών του ευρωπαϊκού σχολείου και επομένως έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το απολυτήριο το ευρωπαϊκό ε, είναι έτοιμα όπως είναι το γερμανικό σχολείο ή το αμερικάνικο σχολείο ή το γαλλικό σχολείο ή πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή προκειμένου να προσαρμοστούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αν το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Σχολείου ε, πραγματικά διεισδύσει στα συστήματα των, ευρωπαϊκών, ε, των, εθνικών, ε, ε, ε, των εθνικών κρατών μελών, γιατί έτσι μόνο νομίζω ότι θα υποστηρίξουν και την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Επομένως, μία ερώτηση, με ποιο τρόπο τα εθνικά σχολεία μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να δίνουν ευρωπαϊκό απολυτήριο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε. Χάνο, Χάνο Τάκουλα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου στις ευχαριστίες που εκφράστηκαν προς τον κύριο Καβαδά από συναδέλφους. Είναι μια πολύ σε βάθος αποτελεσματική ενδελεχής ε, μελέτη αυτή. Κατανοούμε όλοι ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία το θέμα είναι και πρόκειται για το πραγματικά να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα και συνάφεια αφενός για τους ίδιους τους μαθητές, αφετέρου για την διασφάλιση διδασκαλίας στη γλώσσα τους. Αυτό είναι μια ξεχωριστή α, αυτοτελής αξία, η αξία. Όσον αφορά τώρα αυτά τα θέματα, είναι μια ανησυχία που εκφράζουμε. Οι μικρέ γλώσσε πρέπει να διασφαλιστούν και να συνεχίσουν να υφίστανται. Το επεσήμανε αυτό ο κύριο Καβαδά. Όμω, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει ιδιαίτερα να, γίνει, να, να προσέξουμε ώστε οι μικρές γλώσσες να μην απομονωθούν και μείνουν στο περιθώριο. Πιστεύω ότι είναι η βιτρίνα ακριβώς ε, η εικόνα της Ευρώπης που δίνουμε και πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να δίνεται αυτή. Γίνεται λόγος για ε, δυνατότητες ε, που πρέπει να δοθούν τα μικρά παιδιά που μπορούν να συμμετέχουν Πρέπει να δούμε το ότι δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται την υποστήριξη στη μητρική τους γλώσσα. Πρέπει στη μητρική τους γλώσσα αυτά τα μικρά παιδιά να εκπαιδεύονται και να δυνα... γίνεται, δίνεται η δυνατότητα, η κινητικότητα να διασφαλίζεται υπό τις καλύτερες πτυχές. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καβαντά για την εξαιρετική του δουλειά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Συνάδελφε Καβαντά, με έκπληξη έπρεπε να διαπιστώσω ότι πάλι υπό το σημείο 2 διαρωτάστε πρέπει να ζητήσετε, όχι μια στιγμή, μια στιγμή να το ξαναβρω, εδώ, εδώ υπό το σημείο 23 είναι αυτό. Λοιπόν, υπό το 23. Λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο πτυχίο σε χαμηλότερο επίπεδο κάτω από το ακαδημαϊκό απολυτήριο. Εμείς το είχαμε στην τελευταία ή πρώτα τελευταία τουλάχιστον έκθεσή μας το ίδιο αίτημα από πλευρά συναδέφου Περί που είχε συντάξει η έκθεση είχαμε ζητήσει από τα σχολεία και είχαμε πει δεν είναι δυνατόν μόνο με το ακαδημαϊκό απολυτήριο, με το δίπλωμα να μπορούν να αποχωρήσουν οι μαθητές. Πρέπει ενδιάμεσα να υπάρχει κάποιο <clears throat> κατώτερο, χαμηλότερο δίπλωμα, αν δεν φτάσουν ως την τελευταία τάξη, ώστε να διασφαλίζονται αυτά τα παιδιά. Κάτι σαν το Mittlerer Reife στη Γερμανία. Ένα δευτερεύον, θα έλεγα, ε, επαγγελματικής ε, κατάρτισης ε, δίπλωμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, παρατηρούν και γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στου γονεί όταν πρόωρα εγκαταλείπουν το σχολείο. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το σημείο. Το 23 είναι σημείο κλειδί. Δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Θα έπρεπε και θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν περισσότεροι άνθρωποι είχαν πάρει σοβαρά τα αιτήματά μα και τι εκθέσει μα. Κύριε Καβαντά, επιθυμώ η έκθεσή μα να ληφθεί ιδιαίτερα στα σοβαρά και εύχομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να κινητοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Χάνιμπαλ, παρακαλώ, θέλατε η κυρία Χάνιμπαλ. Ευχαριστώ. Και εγώ ήμουν εισηγήτρια για αυτό το θέμα δύο φορές μάλιστα και έτσι τα έχω εξετάσει αυτά τα ζητήματα λεπτομερώς. Εμένα μου φαίνεται ότι δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου από το που έγραψα από τη δική μου έκθεση ε, πριν μερικά χρόνια. Ε, θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ στα σοβαρά. Λοιπόν, συγκεκριμένα τον αριθμό ε, των μελών του προσωπικού, η, η ζήτηση αυξάνεται, δεν μειώνεται. Και έτσι είναι ακόμα πιο σημαντικό να βρούμε ένα σύστημα που να λειτουργεί, γιατί τώρα δεν λειτουργεί. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ε, το, τον σκοπό, το νόημα αυτών των ευρωπαϊκών σχολείων, ποιο θα πηγαίνει σε αυτά τα σχολεία. Γιατί μάλλον ε, φαίνεται σαν να γίνεται μετά από κλήρωση. Και ιδιαίτερα με ε, απασχολεί αυτό που συμβαίνει με την ε, εκπαίδευση, ε, τη διδασκαλία των γλωσσών. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της ε, πρόσληψη ε, δασκάλων. Ήταν δύσκολο πάντα αυτό το ζήτημα. Πάντα ήθιστε να προσλαμβάνονται από τα κράτη-μέλη. Το, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Τα κράτη-μέλη έχουν τους δικούς τους τρόπους να το κάνουν. Όταν εγώ το έκανα αυτό, υπήρχε έλλειψη καθηγητών που δίδασκαν αγγλικά, γιατί το σύστημα στην Αγγλία και την Ουαλία, γιατί στη Σκοτία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το σύστημα λοιπόν εκεί το, χειρίζονται, το οι τοπικές αρχές. Έτσι μπορούν να υπάρχουν παρόμοια εμπόδια και σε άλλα κράτη-μέλη. Όταν λοιπόν κοιτάζουμε την πρόσληψη, σε θεωρητικό επίπεδο όλα είναι καλά. Αλλά δεν ξέρω στην πράξη πώς αυτό λειτουργεί. Και αν μπορούμε να βρούμε καθηγητές με το κατάλληλο επίπεδο. Το διδακτικό προσωπικό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερέστερα για να ε, παρέχουμε διδασκαλία με την κατάλληλο επίπεδο ποιότητα. Και πάλι να υπενθυμίσω κάτι από την έκθεση περί 2002 ή την έκθεση Hannibal 2005 που και στις δύο εκθέσεις υπήρχε αυτό το αίτημα και τι δύο φορέ δεν, την πήραν, δεν το πήραν στα σοβαρά αυτό το αίτημα. Δεν το βρίσκω ιδιαίτερα ευγενικό αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει ευήκο νου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από του αρμόδιου εκεί. επιτέλου, να προβληματιστούν και να σκεφτούν. Δεν θα ήταν καλύτερο να έχουν καλύτερε επαφέ που θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέτοιου είδου σημαντικά ε, αιτήματα του Ευρωκοινοβουλίου να τύχουν συνέχεια. σω μπορεί να απαντήσει εκπρόσωπο τη Επιτροπή, τώρα ο κύριο Μπόρι, και μετά εσεί. Συνάδελφε Μπόρις, έχετε τον λόγο. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου στα συγχαρητήρια προς τον κύριο Καβαντά. Και για το γεγονός ότι σήμερα διοργάνωσε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα ως εκδήλωση. Το θέμα των ευρωπαϊκών σχολείων το έχετε πραγματικά σε βάθος εξετάσει. Ο σημερινός αριθμός των ευρωπαϊκών σχολείων και εξού και ο σημερινός αριθμός των μαθητών απορρέει αποκλειστικά από το ύψος των κονδυλίων του προϋπολογισμού που διατίθεται για τα ευρωπαϊκά σχολεία από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και από τι εισφορέ των κρατών μελών, ή το καταφέρετε να βρείτε τι πραγματικέ ανάγκε που θα αντανακλώνται και να τι διαγνώσετε τι πραγματικέ ανάγκε από αυτή την εικόνα όπω υπάρχει σήμερα. Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων έχουν την ανάγκη μέσω της κινητικότητας μια και ανοίγονται διαρκώς περισσότερες αγορές εργασίας οι ροές οι μεταναστευτικές εντείνονται όλο και περισσότερο προς την Ευρώπη και δεν συνδέονται μόνο με το Λουξεμβούργο εκεί όπου υπάρχουν ισχυρέ έδρες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάποιες πληροφορίες λοιπόν για τις πραγματικές ανάγκες που υφίστανται την πραγματική ανάγκη συνολικά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά σχολεία που θα έπρεπε να καλυφθεί. Καλό θα ήταν να εντείνουμε αυτά τα στοιχεία στην έκθεση και ένα μέρος των κρατών μελών να πούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τους και πρέπει να συγχρηματοδοτούν και να αποστέλουν καθηγητές και διδασκάλους σε αυτά τα σχολεία, αυτά τα κράτη να μεριμνούν γι' αυτό. Θα έπρεπε με σαφήνεια κάθετα να αναφέρεται στην έκθεσή μας αυτό. Αυτό είναι ένα από τα κύρια προβλήματα πιστεύω. Και θα έλεγα και το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο επιπλέον. Πολύ σαφώς, με μεγάλη σαφήνεια το αναφέρεται αυτό. Τα εθνικά συστήματα είναι καμιά φορά, πολλές φορές ασύμβατα με, μεταξύ του. Και είτε μαθαίνουν, ε, εκπαιδεύονται σε γενικά ιστορικά μαθήματα οι μαθητές και μετά όταν έρχεται η ώρα να πάνε για το απολυτήριο έχουν ερωτήματα για την εθνική τους, εθνική τους ιστορία. Για τις εξετάσεις για πανεπιστήμια, για πρόσβαση σε πανεπιστήμια, οι χώρες το απαιτούν αυτό. Θα πρέπει λοιπόν με σαφήνεια να πούμε ότι ένα ευρωπαϊκό απολυτήριο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες πρόσβασης σε όλα τα πανεπιστήμια πανευρωπαϊκά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε για την έκθεση. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Ουμπέρτο Μόρικα από την Επιτροπή παρακαλώ θα έχει τον λόγο. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Euh, Να ευχαριστήσω τον κύριο Καβαντά που μας ε, παρουσίασε την έκθεσή του. Έλα βέβαια και γνωμοδότηση και άλλων επιτροπών, Επιτροπή Προπολογισμού και Δικαστικών Υποθέσεων του ε, Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, κάνει, έχει υποβάλει τις παρατηρήσεις της σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια ενός χειρού τραπέζης προς τον κύριο Καβαντά σχετικά με το σχέδιο έκθεσης. Ε, κάτι το οποίο η Επιτροπή δέχεται ε, με πολύ θετικό πνεύμα σε ό,τι αφορά την ανάλυση αλλά και τα αποτελέσματά της. Για τα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν και συγκεκριμένα το πρόβλημα των ε, πτυχίων ε, που παρέχονται από ε, τα σχολεία, μπακαλαιογεά ή άλλα πιστοποιητικά, αλλά και το ζήτημα της πρόσληψης καθηγητών για το απολυτήριο. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για μια επιτυχία. Υπάρχουν βέβαια στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης, αλλά κυρίως μιλάμε για αξιοποίηση ορισμένων στοιχείων ή, ή για την χρήση των βαθμών μάλλον, για την εισαγωγή μετά σε άλλα σχολεία, σε άλλα κράτη-μέλη. Ε, ε, κυρίως εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα και βεβαίως εργαζόμαστε επ' αυτού. Ε, η Επιτροπή και ο Αντιπρόεδρος Σεφκοβιτς έκανε μια παρέμβαση την προηγούμενη Παρασκευή στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας ακριβώς για αυτό το σημείο και περνώντας τώρα στο επόμενο ζήτημα, ε, για την απόσπαση καθηγητών στα ε, ευρωπαϊκά σχολεία. Υπάρχουν ε, θέσεις που δεν καλύπτονται από καθηγητές που αποστέλλονται από τα κράτη-μέλη. Ήταν ένα σημαντικό, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για δύο λόγους. Πρώτον, από δημοσιονομική πλευράς υπάρχει ένα ζήτημα πόρων, έλλειψη πόρων μάλλον. Αλλά ένα άλλο πιο φιλοσοφικό μάλλον πρόβλημα, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία ε, βρίσκονται ανάμεσα στο, στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα. Η απόσπαση καθηγητών έχει ως στόχο να μεταφέρει στοιχεία από το, από το ένα σύστημα στο άλλο και έτσι να υπάρξει μια σύγκληση μεταξύ των δύο. Βεβαίως γίνονται και διμερείς επαφές ε, με τα κρατη σχετικά με την ε, απόσπαση των καθηγητών. Ούτως ώστε να γίνεται αυτό με τις, ε, υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. και για να βοηθήσουμε αυτά τα κράτη-μέλη. Υπάρχει, πρέπει να πω, και ένα γενικό ε, πρόβλημα σε ό,τι αφορά την απόσπαση των ε, καθηγητών. Μια πολύ ισχυρή ζήτηση, υψηλή ζήτηση για τους αγγλόφωνους καθηγητές, ε, ιδιαίτερα λέει δηλαδή, τους Βρετανούς και τους Ιρλανδούς καθηγητές, και η ζήτηση αυτή υπερβαίνει τον, το ύψος των ε, συνεισφορών που είναι διατεθειμένα αυτά τα κράτη-μέλη να ε, παράσχουν. Υπάρχουν δηλαδή κράτη-μέλη τα οποία κάνουν ήδη αρκετά και πάνω ε, και πέρα από, το, από αυτό που τους αναλογεί. Για την δημιουργία ενός επιστοποιητικού, ενός απολυτηρίου. Ε, για κάποιον που θέλει να στραφεί προς ε, ε, την επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό εμείς θα το παρουσιάσουμε στο Ανώτατο Συμβούλιο την επόμενη φορά για να μπορέσει να συζητηθεί εκεί. Και πρέπει να Βεβαίω, να λαμβάνουμε υπόψη ότι εμεί έχουμε μία ψήφο ω επιστροφή, ω επιτροπή, συγγνώμη, έχουμε μία ψήφο εκεί. Γι' αυτό και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, συμμετάσχουν στο δυνατόν περισσότερο μαζί με την Επιτροπή σε αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε. Η απάντηση φυσικά δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, εντάξει. Το 2002 το ζητήσαμε το 2005 το ξαναζητήσαμε και λέτε 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει θα υποβάλει μια πρόταση. Ε, πώς γίνεται αυτό. Τι να κάνουμε με όλα αυτά που μας είπατε. Καθυστερήσατε πολύ. Μια σαφή εντολή δώσαμε. Τώρα δίνουμε για τρίτη φορά το αίτημα αυτό ως εντολή. Το πρόβλημα της, ε, ε, της πρώιμης αποχώρησης μαθητών από τα σχολεία να αποσαφινιστεί και να δίνεται μια λύση, ένα δίπλωμα ενδιάμεσο για την επαγγελματική κατάρτιση. Τι, ποια δυσκολία υπάρχει, γιατί δεν γίνεται αυτό, αφού γίνεται και σε άλλα σχολεία. Δεν ευθύνεστε, λέει εσεί, αλλά είσαστε εσεί ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μια και είσαστε σύνδεσμό μα εσεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να ενδιαφερθείτε γι' αυτό. Δεν είναι σωστό, είναι απαράδεκτο. Και θα έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια να είχαν υπάρξει επερωτήσεις και να είχαν αποσαφινιστεί αυτά. Δεν μπορώ εγώ, δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνη, ο υπεύθυνο εφόλων αυτών και με κάθε σοβαρότητα. Παρακαλώ εξ ονόματο όλων των συναδέλφων να μεριμνήσετε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόβλημα των πρώιμων αποχωρήσεων από την, ε, τα ευρωπαϊκά σχολεία να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα άλλα τα οποία συνεπάγεται αυτό επιτέλους στα ευρωπαϊκά σχολεία να ληφθεί αυτό υπόψη και όχι μόνο σε σχέση με τα κράτη-μέλη ή τα εθνικά συστήματα που δεν έχει καμιά αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λέτε θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση και να μειωθεί ο αριθμό. Εκεί που έχετε εσεί όμω αρμοδιότητε δεν κάνετε τίποτα. Εντάξει, λοιπόν, με κάθε ευγένεια το ζητώ. Κυρίε κύριοι, να το λάβετε αυτό με σοβαρότητα υπόψη και να το αποσαφηνήσετε. Και παρακαλώ του συναδέλφου να μεριμνήσουν σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία να τύχει συνέχεια σε αυτό το θέμα και να το προωθήσουμε. Θα σα ξαναρωτήσουμε το φθινόπωρο. Το κάνατε ή όχι. Και κάθε κάθε εποχή, κάθε, ε, εποχή του χρόνου θα ρωτάμε αν το κάνατε ή όχι. Και θα ρωτάμε, κάνατε τη δουλειά σας ή όχι, όπως οι δάσκαλοι τους μαθητές. Ο κύριος Καβαντά λοιπόν έχει τον λόγο, παρακαλώ. Θέλετε να παρέμβετε εσείς ή όχι. Euh, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Εσείς η οχι οπως οι δασκαλοι τους μαθητες ο κυριος καβαντα λοιπον εχει τον λογο παρακαλω θελετε να παρεμβετε εσεις η οχι θα ειμαι παρα πολυ συντομος προεδρε εσεις οι ιδια θεμητά εκνευρισμένη μετά από εννέα χρόνια ενός αμαξιδίου το οποίο θα πρέπει να σπρώχνουμε σε μία μόνιμη ανηφόρα είναι κάτι το οποίο εξαντλεί. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις κρίσεις τους και τις αναλύσεις τους. Είμαστε στη διάθεσή τους για να μπορέσουμε να δεχθούμε μέσω των τροπολογιών τους ότι έχουν να προτείνουν. Καταλήγοντας θα ήθελα να θέσω δύο θέματα. Το πρώτο αφορά τις βασικές αρχές και το δεύτερο αφορά τα μέσα. Σε επίπεδο αρχών, να θυμίσω ότι στόχος αυτών των ευρωπαϊκών σχολείων δεν είναι να είναι ένα τελικό συμπλήρωμα μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε το προσωπικό που δουλεύει στα ευρωπαϊκά όργανα. Καταρχάς το προσωπικό των ε, οργάνων, το οποίο θεωρείται ευνοημένο γιατί έχει τέτοιου είδους σχολεία που οι περισσότεροι βάζουν τα παιδιά τους, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να ασκούν το δικαίωμά τους. Σήμερα το πρωί υπήρχαν αναφορές και σε προσωπικό που εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 1.600 ευρώ το μήνα. Δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Αν δούλευαν στην πατρίδα τους τότε το σχολείο τους θα ήταν δωρεάν για τα παιδιά τους. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί τα θεσμικά όργανα θα αρνηθούν να αναλάβουν αυτήν τη συγκεκριμένη υποχρέωση η οποία θα έλεγα είναι το λιγότερο που προσφέρουν σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σαν παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό το μέσο που έχουμε, αυτό το πράγμα που υπάρχει και έχουμε στη διάθεσή μας, δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να χαθεί. Δεύτερον, τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν είναι μόνο ένας χώρος ο οποίος απλά βοηθά τις οικογένειες να τοποθετούν τα παιδιά τους και στα θεσμικά όργανα. Είναι ένας χώρος όπου θα έλεγα ασκείται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξ αρχής, με πολλές γνωσικές γνώσεις, με πολιτισμικές, πολυπολιτισμικές επαφές και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα τη στιγμή κατά την οποία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο εθνικισμός που είναι ο προθάλαμος πολλών άλλων δυσκολιών αντιμετωπίζει νικηφόρα τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πολιτικής και νομίζω ότι δεν πρέπει να αγνοούμε μόνο τα παιδιά, ε, μάλλον δεν πρέπει να αναφερόμεθα μόνο στα παιδιά του προσωπικού γιατί υπάρχουν παιδιά και άλλων πολιτών που βρίσκονται στις συγκεκριμένες πόλεις όπου λειτουργούν τα σχολεία. Τώρα λοιπόν για τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους τα σχολεία. Υπάρχουν προβλήματα για τους πόρους των σχολείων και για τον προϋπολογισμό. Η Επιτροπή κάνει μια προσπάθεια. Θα πρέπει όμως να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο να δίνει περισσότερα κίνητρα και να υποχρεώνει λίγο τις χώρες που δεν σέβονται τις υποχρεώσεις τους, είτε σε καθηγητές είτε σε χρήματα. <clears throat> Κατανοώ ότι οι Βρετανοί δεν είναι πολύ, εν δεν είναι σε πολύ εύκολη θέση, γιατί όλοι θέλουν να μιλούν την αγγλική γλώσσα, αλλά σε ένα κοινοτικό σύστημα, όταν κάποιος δίνει πολλά παίρνει περισσότερα, οπότε Τέλος. Είπατε κυρία Πακ κάτι το οποίο εκπλήσει. Αν χρειάζονται εννέα χρόνια για να μετακινηθεί έστω κατά κάποια εκατοστά ένα σύστημα, αυτό σημαίνει ότι το εκτελεστικό δεν ήταν στο επίπεδο της αποστολής του. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι από ότι αυτά τα 20.000 άτομα που καλύπτονται. Βρισκόμαστε επίσης σε ένα συσχετικό θα έλεγα δυνάμεων ο οποίος λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστή, σαν καύσιμο. Να δημιουργήσουμε λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί μαζί με τους προσκεκλημένους που είχαμε το πρωί στη Στρογγύλη Τράπεζα τα πράγματα, να ελέγχει τα πράγματα και να τροφοδοτεί θα έλεγα την προσπάθεια που κάνουμε. Δεν κάνουμε πολιτική στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ μιλάμε για την εκπαίδευση. Δεν θα σας θυμίσω αυτά που είπε ο ότι αν ήταν να ξεκινήσω εκ νέου την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινούσα από την εκπαίδευση αυτή τη φορά. Ναι. Άλλοι λένε ότι το είπε ότι θα ξεκινήσω με τον πολιτισμό αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ξεκίνησε με την οικονομία, χωρίς να ξεχνά βέβαια τον πολιτισμό και την παιδεία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καβαντά. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης. 14 Ιουνίου, καταληκτική προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. 24 Ιουνίου, εντάξει, καταληκτική προθεσμία για τις τροπολογίες. 13-14 Ιουλίου ψήφιση για έγκριση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ελπίζουμε στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ήδη τώρα να ξεκινήσει τη δουλειά της. Δεν χρειάζεται να εγκριθεί στην Ολομέλεια πρώτα για να συνεχίσει. Μπορείτε ήδη τώρα να ξεκινήσετε με την εργασία σας προς αυτήν την κατεύθυνση. Εντάξει, συμφωνείτε. Τέλεια. Λοιπόν, σημείο 5 της ημερησίας διάταξης τώρα. Η ημερήσια διάταξη για δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Έχουμε μια πρωτοβουλία ναυαρχίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που έχει αναλυθεί για το 2020 είναι η απασχολησιμότητα αυτή η ναυαρχίδα. Και φυσικά η συνάδελφος ε, κυρία ε, Νεβίδα Λόβα έχει αναλάβει την ε, έκθεση αυτή. Θα μας την παρουσιάσει τώρα. Παρακαλώ κυρία Νεβίδα Λόβα. Καταρίνα έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το ποσοστό ανέργων στους νέους είναι 21,4% πολύ υψηλό. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός. Υπάρχουν όμως χώρες όπου προσεγγίζει το ποσοστό αυτό το 40%. Χαιρόμαστε ότι στην ημερήσια διάταξη 2020, στη στρατηγική για το 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εγγραφεί αυτό το πρόγραμμα νέων συγκεκριμένων εξειδικευμένων δεξιοτήτων για νέε θέσει απασχόληση. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του σκιώδει εισηγητέ, με του οποίου είχαμε πολύ καλέ επικοδομητικέ συζητήσει και επαφέ. Βρισκόμαστε, α το πω έτσι, όλοι σε, ως επιβάτες στο ίδιο πλοίο, στο ίδιο σκάφος. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η γνωμοδότηση που είναι σύντομη και περιεκτική. Ελπίζω ότι όλοι την έχουν διαβάσει. Υπάρχουν κάποια σημεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ούτως ή άλλως υποστηρίζουμε τις δεξιότητες εκείνες που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για το μέλλον. Γλωσσικές δεξιότητες και προσόντα, παράδειγμα, επιπλέον πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες που οι πολίτες μας στο μέλλον θα χρειάζονται ιδιαίτερα για να προχωρήσουν η Ευρώπη. Σε αυτή την πρόταση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων στην εκπαίδευση των εργοδοτών, των Υπουργείων στα επιμέρους κράτη-μέλη θα πρέπει να ενταχθεί, να ενταχθεί. Είναι σημαντικός αυτός ο παράγοντας ώστε να δημιουργηθεί μια εικόνα εκείνου που παίρνει πτυχίο από την σχολική εκπαίδευση διπλωματούχου για να μπορέσουμε να καθορίσουμε ποια θα είναι η εικόνα αυτού του προσοντούχου νέου. Πολύ σημαντικό αυτό, να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα εμπεριέχεται στα συστήματα τα εκπαιδευτικά, τι θα προσφέρετε στους νέους ως γνώση. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία θέλουμε, θέλω να υποστηρίξω με κάθε τρόπο σε αυτό το πλαίσιο. Πολύ σημαντικό είναι και η άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση και η αναγνώριση αυτής της εντός εισαγωγικών άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Να φανταστείτε το έργο αυτό που πρέπει να επιτελεστεί και σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν άτυπες τέτοιες ικανότητες και δεξιότητες που πολύ σπάνια σήμερα αναγνωρίζονται. Είναι, ας το πω έτσι, μια πρόσθετη αξία αυτή που χρειάζονται όλοι. Πρέπει να υπάρχει ένα εξειδικευμένο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα ονομάζεται για παράδειγμα Λεωνάρντο Νταβίντσι για να υποστηριχθούν οι νέοι. Χρειάζεται χρηματοοικονομική υποστήριξη για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει βιώματα και εμπειρίες, ώστε με εξειδικευμένη κατάρτιση και απόκτηση γνώσεων να αποκτήσουν οι νέοι την κινητικότητα εκείνη που απαιτείται, ώστε να μπορέσουν να βρουν απασχόληση στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισή του και να μπορούν να εκπαιδευτούν και στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε όλα να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα Έρασμος. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και πρέπει να συνεχιστούν. Έχουμε προγράμματα όπως οι νέοι σε κινητικότητα ή η κινητοποίηση σε σχέση με τη νεολαία και παρακαλούμε αυτά τα προγράμματα να τύχουν υποστήριξης. Δυστυχώς μόνο 20 λεπτά έχω στη διάθεσή μου. Όμως θα ήθελα να δώσω ευκαιρία στους συναδέφους να τοποθετηθούν σε αυτά τα θέματα και έτσι ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Χάνου Τάκολα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάκολα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Tässä osaltani lausun kiitoksia myös meidän. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας και ε, επίση και την κυρία Μονέσκου η οποία με βοήθησε πάρα πολύ για να διαμορφώσω μια εμπεριστατωμένη άποψη γύρω από αυτήν την καλή θα έλεγα έκθεση. Νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία υπογραμμίζει έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Καταρχάς, προφανώς και πρέπει να υποστηρίξουμε με καλύτερους οικονομικούς πόρους στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Αυτή είναι, αυτός είναι ο στόχος μας για το πρόγραμμα του 2020. Από την άλλη, αυτό το οποίο μας απασχολεί στη συγκεκριμένη φάση είναι να μπορέσουμε να βρούμε ε, πιο ευέλικτες λύσεις έτσι ώστε η εκπαίδευση και η κατάρτιση να μπορέσουν να καλύψουν καλύτερα από ό,τι το κάνουν σήμερα τις ανάγκες της αγοράς. Έχουμε, θα έλεγα, μια ευρωπαϊκή προοπτική εδώ και σε πλαίσια αυτή της προοπτικής θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις μεγαλύτερε επιχειρήσεις. Αυτό είναι προ το συμφέρον όλων. και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον ακαδημαϊκό χώρο και τα πανεπιστήμια τα οποία θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο από ό,τι σήμερα. Αυτό εν πολλής θα έλεγε κανείς ότι συμβαίνει σε ορισμένες τουλάχιστον χώρες μέλη. Αλλά δεν είναι γενική η διαπίστωση αυτή. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα καλό πρόγραμμα. Και είμαστε και ικανοποιημένοι και από τις προτάσεις της κυρίας Νεβέλοβα. Συνάδελφος Λότα Μπίσκι παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση πιστεύω. Μια σκέψη θα ήθελα να εκφράσω που θα μπορούσε να υπογραμμιστεί ακόμα πιο πολύ. Πρόκειται για την ανάγκη της παραδόσης ε, των ε, χειρονακτικών επαγγελμάτων ως δεξιότητες να τις διασφαλίσουμε στην επιβίωσή τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αυτά τα επαγγέλματα να διασφαλιστούν να μην εξαφανιστούν, μια και απειλούνται με εξαφάνιση. Για παράδειγμα, η παράδοση των, ε, της δημιουργίας ε, καλών φρακτών από χειρόνακτες. Εξαφανίζονται όλα αυτά. Βιομηχανικά παράγονται και είναι το ίδιο προϊόν τυποποιημένο. Κρίμα είναι. Όταν έχουμε καλλιτεχνικές βιοτεχνίες ε, και χειρονακτικές εργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να καλλιεργηθούν και να διασφαλιστούν εν μέρη δεν υπάρχει δυνατότητα να εκπαιδεύονται όπως πρέπει αυτοί που θέλουν να μάθουν για παράδειγμα να ασχοληθούν ως με τη σφυριλασία των μετάλλων να μπορούν να δημιουργούν αυτά τα καλλιτεχνήματα. Κρίμα θα ήταν γιατί θα έχανε η Ευρώπη έτσι ένα σημαντικό πολιτισμικό κληροδότημα που έχει. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο κύριος Φίσας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην κυρία Νέντελα Λόβα για την έκθεση που συνέταξε που θεωρώ ότι είναι περιεκτική και πλήρης. Θα ήθελα να σχολιάσω δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα και είναι ιδιαίτερο μέλημα και ανησυχία δική μου υποστήριξη στην επαγγελματική κατάτηση. Στη σημερινή συγκυρία είναι πολύ σημαντικό αυτό και ιδιαίτερα ο τρόπο να το αναβαθμίσουμε. Να μην είναι δεύτερη κατηγορία η επαγγελματική κατάτηση ή κάτι το, το οποίο δεν είναι άξιο ε, να αναγνωριστεί και να αξιολογηθεί όπω είναι το επάγγελμα των ιατρών ή των μηχανολόγων ή μηχανικών. Είναι πολύ σημαντικό τα επαγγέλματα αυτά η κατάρτισή τους να μην είναι δεύτερο, δεύτερου επίπεδου, δεύτερης κατηγορίας, να έχουν την ίδια αναγνώριση και κύρος όπως τα άλλα ακαδημαϊκά επαγγέλματα. Και εδώ και το θέμα της ε, απασχόλησης θα έλεγα είναι σημαντικό. Είναι μια σημαντική πηγή δημιουργίας απασχόλησης και πρέπει έτσι να τον αντιμετωπίζουμε. Και με αυτό το οποίο ανέφερε ο συνάδελφος και συμφωνώ απόλυτα με τα βιοτεχνικά επαγγέλματα και τις ε, χειροτεχνικές αυτές ε, ε, ικανότητες θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε μαθητευόμενους να εκμάθουν, να ασχοληθούν και να εξοικειωθούν με αυτές τις δεξιότητες. Αυτού του είδους οι δεξιότητες χειρονακτικών και βιοτεχνικών επαγγελμάτων να μην απολεστεί πολλοί νέοι να έχουν την διασφάλιση ότι θα μπορούν να ασκήσουν αυτά τα επαγγέλματα και έτσι δεν θα χαθούν αυτά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την ε, Καταρίνα για την πλήρη περιεκτική αυτή έκθεση. Θέλω να προσθέσω κάποια θέματα. Είχα την ευκαιρία επί 7 χρόνια να ασχοληθώ με την επαγγελματική κατάρτιση στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Το πρώτο θέμα που θα έπρεπε να αναφέρουμε είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Μπίσκι ο ίδιος πιο πριν. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε την ανεργία να την καταπολεμήσουμε και να τη μειώσουμε την ανεργία των νέων προσφέροντας δυνατότητες να εξοικειωθούν και να καταρτιστούν οι νέοι σε όλα τα επίπεδα σε αυτή την επαγγελματική κατάρτιση. Να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που υπάρχουν ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς, την προσφορά στις αγορές, στις αγοράς. Για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να γίνει σιδηρουργός και να ασχοληθεί με τη σφυριλάτηση τέτοιου είδους ε, ε, ε, καλλιτεχνημάτων ή και στο περιφερειακό τοπικό επίπεδο, εθνικό επίπεδο λιγότερο στο ευρωπαϊκό αλλά στο εθνικό τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Είναι σημαντικό λοιπόν, θα ήταν σημαντικό υπό αυτό το πρίσμα της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την επαγγελματική κατάρτιση υπό το πρίσμα των αναγκών των αγορών της αγοράς, μακροπρόθεσμα να σχεδιάσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες. Επικοδομητικό θα ήταν αυτό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κάποια απόφαση που μπορεί να είναι λανθασμένη από πλευράς κάποιου νέου, όταν ε, επιλέγει κάτι το οποίο δεν έχει κάποια προοπτική και Το είπε η Καταρίνα τον Ιούνιο. Θα συζητήσουμε τα θέματα του νέου προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε συνολικά πώ το, το πρόγραμμα τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση θα διαμορφωθεί το Λεωνάρντο Νταβίντσι Συν αποτελεί ένα μέρο, ένα τμήμα αυτού του προγράμματο. Θα θέλαμε όμω σε αυτή την έκθεση να τονιστεί περισσότερο αυτό, ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να εξετάζεται και να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί υπό το πρίσμα της επαγγελματική κατάρτιση. Και έτσι πρέπει να το εγκρίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το, το πρόγραμμα τη διαβίου εκπαίδευσης και μάθηση και κατάρτιση πρέπει με αυτόν τον τρόπο να στηθεί στα πόδια του. Και με το έρασμο η αύξηση τη δυνατότητα επαγγελματικών ε, ε, δεξιοτήτων και γνώσεων για τους νέους. Ένα πράγμα πρέπει να τονίσουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 100 εκατομμύρια ευρώ. Και ακριβώς ε, γι' αυτό το στόχο χρησιμοποιούνται και πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να μπορέσει να διασφαλιστεί και να διατηρήσει τις δράσεις του που θα στοχεύουν στους νέους. Και το μελλοντικό πρόγραμμα της διαβίου εκπαίδευσης Lifelong Learning από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηριχθεί. Ευχαριστούμε. Κύριε Παπα-Νικολάου, έχετε τώρα εσείς τον λόγο, παρακαλώ. Ε, thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Πράγματι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα κατά αυτή την περίοδο. Είναι μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και βεβαίως ως ε, Επιτροπή Πολιτισμού υποβάλλουμε προτάσεις για να δώσουμε, παράσχουμε περισσότερες δεξιότητες στους νέους για να είναι σε θέση να αποκτήσουν μια καλύτερη, μια καλύτερη δουλειά, μια καλύτερη ζωή στο μέλλον. Κάτι άλλο στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι η ισορροπία που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ ε, ανάμεσα στις δεξιότητες αφενός και στις ε, θέσεις εργασίας που προσφέρονται. Γιατί σε πολλά κράτη-μέλη, συγκεκριμένα αναφέρομαι στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ε, μεγάλες ε, οικονομικές δυσκολίες, οι νέοι εκεί έχουν δεξιότητες, αλλά δεν βρίσκουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας. όπου θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες. Έτσι, με αυτή την απώλεια εγκεφάλων, brain drain, ε, αυτό έχει καταστη... είναι πλέον μια τάση και χάνουμε έτσι ικανούς ανθρώπους, έξυπνους νέους ανθρώπους που ε, προσπαθούν να βρουν, ε, να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή, πολύ πιθανό και σε μια άλλη ήπειρο. Αν λοιπόν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό στο άμεσο μέλλον, Πολύ σύντομα θα είναι αργά. Ευχαριστούμε κύριε Παπα-Νικολάου. Στι πίσω σειρέ ε, έχουμε το εμπορικό επιμελητήριο από τον Νότιο Τυρόλο υπό την πρωτοκαθεδρία ε, συναδέλφου μας ε, που ήρθαν εδώ. Καλώς ήρθατε Καλώ ορίσατε. Συζητάμε τη νέα ημερήσια διάταξη για νέε θέσει απασχόληση και νέε κατευθύνσει μέχρι το 2020. Είναι ένα θέμα που και στη δική σα εκλογική περιφέρεια σίγουρα συζητείτε. Σα ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι θα μπορέσετε να δείτε πραγματικά ότι οι ευρωβουλευτέ κάνουν κάτι το θετικό εδώ. Μην πιστεύετε του δημοσιογράφου. Ε, που σας λένε κάποιες ανοησίες. Εδώ γίνεται καλή δουλειά και πάλι καλώς ορίσατε θερμά. Επανέρχομαι στο θέμα αυτό και θα ήθελα να ανταποκριθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Μπίς και ο κύριος Παπα-Νικολάου και ο κύριος Μπόρης και να τοποθετηθώ. Αν δούμε κάτι, την Ισπανία, την Ελλάδα, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο υψηλό ποσοστό νέων ανέργων πρέπει να διαρωτηθούμε ποια είναι τα αίτια, πού βρίσκονται τα προβλήματα, ποια είναι τα λάθη. Γιατί συμβαίνει αυτό έτσι εκεί και όχι στη δική μας χώρα ή στη δική μας περιφέρεια. Στη δική μου περιφέρεια δεν υπάρχει τέτοια υψηλή, τέτοιο υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων. Δεν θέλω να πω ότι είμαστε οι καλύτεροι, αλλά έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα. Πάντα πιστεύαμε ότι η Ευρώπη υπάρχει ώστε να μαθαίνουν οι χώρε από τι βέλτιστε πρακτικέ των άλλων. Έχουμε ένα διοικό, διτό σύστημα. Όχι μόνο εμεί στη Γερμανία, αλλά και στην Αυστρία, στην Ολλανδία. Έχουμε ένα διτό σύστημα όπου η κατάρτιση γίνεται και στι επιχειρήσει και στα σχολεία όμως και οι επιχειρήσεις ε, και η βιομηχανική αυτή δυνατότητα απουσιάζει λύπη όπως είπε ο κύριος Μπίσκι. Πρέπει να μεριμνήσουμε η αγορά εργασίας να είναι πιο διαφοροποιημένη. Να μην έχουμε μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, να υπάρχουν και μικρές επιχειρήσεις. Πολλές μικρές επιχειρήσεις που θα προάγουν τα ταλέντα, του ταλαντούχους νέους, προσοντούχους νέους όπως θα πρέπει. Και να μην έχουμε ένα ισοπεδωτικό σύστημα ώστε να είναι κανεί υποχρεωμένο ε, να πηγαίνει υποχρεωτικά σε ένα σχολείο, αλλά να μπορεί στα 14 να παίρνει ένα πτυχίο από το σχολείο, ένα ενδιάμεσο δίπλωμα, να πηγαίνει στην επαγγελματική κατάρτιση, εκεί να ολοκληρώνει τι δεξιότητε και τι ικανότητε του για να βρίσκει μια δουλειά. Υπάρχουν βέλτιστε πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν το πρόβλημα στην Ελλάδα, τα προβλήματα στην Ελλάδα και τα προβλήματα στην Ισπανία και αλλού να αντιμετωπιστούν όπω πρέπει, με καλύτερο τρόπο. Κρίμα ότι τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργήσαν αυτά τα πράγματα δεν συζητήθηκαν και δεν προχώρησαν όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες βρίσκω και πιστεύω η ανεργία των νέων που είναι μάστιγα της ανθρωπότητας να αντιμετωπιστεί και να αναχαιτιστεί, να σταματήσει. Και πρέπει γιατί αυτή η ατζέντα, η μερίσια διάταξη για δημιουργία θέσεων απασχόλησης με δεξιότητες είναι σημαντική υπόθεση. Αυτά που είπε η συνάδελφο Νέντελα Λόβα και ο κύριο Μπόρι είναι και αυτά σημαντικά. Πρέπει να μεριμνήσουμε τα νέα προγράμματα και μέσω των προϋπολογισμών και των κονδυλίων για αυτά τα νέα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα να έχουν νόημα και να μπορέσουν να έχουν σάρκα και οστά και να συνεχίσουν να υφίστανται, να διατηρηθούν. Θα ήθελα να πω ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω θα το διαβιβάσετε προς τους αρμοδίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το καταφέραμε να παρακολουθεί το πρόγραμμα νεότητας σε κινητικότητα. Διότι ξέρουμε ότι τα προγράμματα που έχουμε είναι φάρη και έχουν έτσι εγκριθεί. Και τώρα να έρθει εκ των όπισθεν κάτι και να έχουμε ένα σύννεφο ε, φεστιακή ε, στάχτης και θάλης ε, που όλα αυτά θα τα συγκαλύψει και θα δοθεί ένα νέο, ένα νέο όνομα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είναι σκληρή μάχη από τον Ιούνιο και πέρα, ώστε να εξευρεθεί ο καλύτερος δρόμος, η καλύτερη πορεία για τα νέα προγράμματα. Παρακαλώ να μην παγιδευτείτε, να μην καταλήξετε στο πουθενά. Όταν έχουμε μια νέα ημερήσια διάταξη για θέσει απασχόληση, τα θετικά αυτά που δημιουργήσαμε και έχουμε ω ναυαρχίδε πρέπει να τύχουν συνέχεια και να διατηρηθούν και να μην ε, οπισθοδρομήσουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό και μπορούμε έτσι νομίζω να επωφεληθούμε. Υπάρχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να παρέμβει. Εσείς κύριε Λεμπραν, είσαστε παρόν. Θέλετε να παρέμβετε. Δεν παρίστατε. Ο κύριος. Ο κύριος Ουμπέρ ή Χούμπερ είναι εδώ. Παρακαλώ. Εδώ είναι, ναι. Ευχαριστώ. Ορισμένες παρατηρήσεις να κάνω. Αρχικά να πω ότι η Επιτροπή συμφωνεί απολύτως ε, με τις ε, προτάσεις ε, της συγγήτριας. Πολύ σωστές μας φαίνονται. Αυτό που εμείς υπογραμμίσαμε στο ε, δικό μας κείμενο, την ατζέντα για τις ε, νέες δεξιότητες και νέες θέσεις απασχόλησης, είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, ε, την επένδυση μάλλον στην εκπαίδευση και κατάρτιση και κυρίως στην τεχνική επαγγελματική κατάρτιση. Δεν πρέπει να θεωρείται ως δεύτερη επιλογή. Ουσιαστικά εμείς υποστηρίζουμε την διοργάνωση του Euroskills, αυτού του διαγωνισμού που θέλει να αναδείξει ε, επαγγέλματα ε, που προκύπτουν μετά από μια τεχνική ε, επαγγελματική κατάρτιση και έτσι αξιοποιούν ορισμένες δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω επαγγελματικής κατάρτισης. Πράγματι, θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα, αυτή την ατζέντα. Έχουμε ε, δρομολογήσει δραστηριότητες ε, για το σκοπό αυτό. Συνέχιση της ανάπτυξης ενός πανοράματος ε, μιας γάμας ευρωπαϊκών δεξιοτήτων για να ε, συλλέγεται το σύνολο των οικονομικών γνώσεων που παράγεται για να ε, αυξήσουμε τα επίπεδα διαφάνειας σε αυτές τις πληροφορίες και σε αυτές τις γνώσεις και πάντα σε διευρωπαϊκό επίπεδο για να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους που δεν βρίσκουν απασχόληση στις χώρες τους ή στις περιφέρειές τους να βρουν μια θέση απασχόλησης κάπου αλλού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ευρωπαϊκό πανόραμα λοιπόν θα μπορούσε να ε, συνεισφέρει σε αυτό το στόχο, αλλά επίσης μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας ανταλλαγής ε, μεταξύ ευρωπαϊκών, ευρωπαίων εμπορογνωμόνων, να υπάρξει μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών λοιπόν. Ένα παράδειγμα πρόσβασης, ε, δράση συγγνώμη, που πάει προς αυτή την κατεύθυνση, δεν ξέρω πώς θέλει να μας πει η συνάδελφος κάτι για την εκπαίδευση. Να προσθέσω μόνο κάτι για όσα υπόθηκαν ε, εδώ. Συγκεκριμένα για το καθεστώς μαθητευομένου. Ε, πρέπει να αποφύγουμε ε, αλληλεπικαλύψεις γιατί υπάρχει ήδη το καθεστώς του ασκουμένου που έχει ήδη προταθεί. Ε, και σε ό,τι αφορά την ε, προώθηση προγραμμάτων όπως το Λουνάρντο Νταβίντσι, βεβαίως ε, και συμφωνούμε. Okay. Μάλιστα, πολύ καλά. Όλες αυτές είναι οι ιδέες που θα συλλέξουμε, συλλέγονται και σημειώνουμε. Είναι όλες αυτές οι ιδέες που εκτίθενται και που μπορούν να συλλεχθούν και θα επηρεάσουν ίσως ιδέες στη συνέχεια μέσα σε αυτό το πλαίσιο να μην ξεχνάμε ότι τα διαθωτικά ταμεία διαδραματίζουν εδώ ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και όχι μόνο το Λεωνάρντο Νταβίντσι. Περισσότερα κονδύλια λοιπόν έτσι μπορούν να διατεθούν και πολλά μπορούν να γίνουν για την κατάσταση Τη διασφάλισης και θέσεων απασχόλησης στις περιφέρειες, στις περιοχές μας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις χειρονακτικά για την ε, μάθηση αυτών των επαγγελμάτων και δεξιοτήτων στους νέους. Πολύ καλά η συνάδελφος Καταρίνα έχει υποβάλει προτάσεις, δεν χρειάζονται πολλέ τροπολογίε. Καταρίνα θέ να ξαναπεί κάτι, να παρέμβει, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που παρενέβησαν, όλους τους προλαλήσαντες και που επεσήμαναν και έδωσαν προσοχή σε αυτά τα προγράμματα. Είναι μεγάλη αυτή η υπόθεση και σε διαφορετικές διασκέψεις που παρακολούθησα και στην Τουρκία ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτή την πρωτοβουλία. Με ικανοποίηση βλέπω ότι εκπροσωπείται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την τελευταία φορά δεν ήταν κανείς παρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν την δυνατότητα υποστήριξης των επιχειρήσεων των βιοτεχνιών επιχειρήσεων. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι και ο κύριος Μπίσκι υποστηρίζει το αίτημα αυτό. Να υπάρχει δυνατότητα εκμάθησης καλλιτεχνικών τέτοιων επαγγελμάτων ως, από πλευράς επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει η κατάρτιση αυτή στα, στα, ε, στα χειροτεχνικά αυτά, βιοτεχνικά επαγγέλματα να ενισχυθεί. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις. Αν υπάρχουν περαιτέρω παρατηρήσεις ευχαρίστως να τις εντάξω στην έκθεσή μου αυτές τις παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία 16 Ιουνίου. Τον Ιούλιο, όπως είπα, θα γίνει Θα ψηφίσουμε. Α, στις 14 Ιουνίου, συγγνώμη, συγγνώμη, 14 Ιουνίου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Τον Ιούλιο θα ψηφίσουμε προ έγκριση στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή. Τώρα επιτρέψτε μου να σα υποβάλω μια πρόταση η κυρία Κώστα βρίσκεται σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Γυναικών. Μπορεί να επανέλθει στη συνέχεια. Το σημείο του συναδέλφου Τάκολα να επισπευστεί λοιπόν. Περνάμε πρώτα στο σημείο 7, προτού γίνει λόγος για το 6. Πάμε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού της Οικονομικής Πολιτικής λοιπόν. Ο Χάνο Τάκουλα. Έχεις τον λόγο Χάνο Τάκουλα, παρακαλώ puheenjohtaja. Στάκουλα, Τάκουλα, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Tämän otsikon taas nähdessäni όταν βλέπω για μια ακόμη φορά το συγκεκριμένο θέμα μπροστά μου, και γνωρίζοντας το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον τομέα της οικονομίας, ε, σκέφτομαι αυτά τα οποία λέει ένας φιλανδός οικονομολόγος, ότι όλοι ομιλούν για την οικονομία και όσο περισσότερο μιλούν τόσο λιγότερο καταλαβαίνουν. Ελπίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ να είμαι σε κάπως καλύτερη κατάσταση. Ελπίζω να έχω καταλάβει κάπως περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη φαίνεται ότι έχουμε στερέψει από γνώμες για την ευρωπαϊκή οικονομία και για τον οικονομικό συντονισμό. Το εξάμεινο δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν πήγε πραγματικά καθόλου καλά στον τομέα του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Εμείς είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις για τον τομέα ο οποίος μας ενδιαφέρει και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ποιοτική εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εξέλιξη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δυστυχώς το θέμα της παιδείας γενικότερα δεν έχει ληφθεί υπόψη στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν περιλαμβάνεται στις 10 κατά προτεραιότητα δράσεις οι οποίες προτείνονται και εδώ θα συμφωνήσω με την πρόεδρό μας, η οποία πριν μερικούς μήνες είχε πει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει λίγο ε, να μην έχει, να μην αγνοεί την ε, εκπαίδευση έτσι όπως το κάνει μέχρι τώρα. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει εκπαιδευμένους πολίτες έτσι ώστε να τονώσει τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, και θα πρέπει η πρόσβαση στην εκπαίδευση να είναι ανοιχτή για όλους. Έχουμε να κάνουμε με μία θα έλεγα έχουμε να κάνουμε με μια αλυσίδα. Το επίπεδο της εκπαίδευσης εξαρτάται από την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι αρμοδιότητες των διδασκόντων σαν παράδειγμα και αυτές εξαρτώνται από την εκπαίδευσή τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά είναι κάτι το οποίο αφορά και τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευόντων έτσι ώστε να πετύχουν τους στόχους τους οποίους θέτουν σε αιτήσια βάση. Πρέπει λοιπόν εμείς να ξεκαθαρίσουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η εκπαίδευση και έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης οικονομικής. Όλες οι μορφές εκπαίδευσης έχουν ε, πολύ μεγάλη σημασία. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, επαγγελματική, επαγγελματική κατάρτιση διαβίου κατάρτιση και παραλαμβάνω είναι πάρα πολύ κρίμα γιατί στις 10 δράσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχει τίποτα για την παιδεία. Γιατί όπως είπαμε η παιδεία είναι κάτι, η εκπαίδευση συγγνώμη είναι κάτι το οποίο λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για πάρα πολλά θέματα στα οποία θέλουμε να προχωρήσουμε. θα πρέπει να έχουμε σαν βασικό στόχο κανένας καταρχάς να μην εγκαταλείπει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Θα πρέπει επίσης να μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποια κοινά κριτήρια για να υπολογίζουμε τα επιτεύγματα και τον βαθμό ικανοποίησης τον οποίο παρέχει η εκπαίδευση στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείπουν τα σχολεία ε, τα ποσοστά των παιδιών που το κάνουν σήμερα. Αυτό το 10% το οποίο για κάποιους θεωρείται ανεκτό είναι ένα στόχος ο οποίος θα πρέπει να ξεπεραστεί. Και τέλος, η βασική έρευνα η οποία στα πανεπιστήμια είναι τα θεμέλια της έρευνας και της ανάπτυξης της οικονομίας, θα πρέπει να αυξηθεί κατά 40% μέχρι το 2020. Φαίνεται ότι στην Ευρώπη αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πετυχαίνουμε μικρά βραχυπρόθεσμα πράγματα, να βάζουμε στόχους οι οποίοι να μην έχουν καμία σχέση με μια μακροπρόθεσμη λογική ανάπτυξης και έρευνας. Πρέπει λοιπόν να αναπροσανατολίσουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπα-Νικολάου, έχετε τον λόγο. Thank Uh, Σε ευχαριστώ και πάλι. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Πάπουλα για το έργο που επετέλεσε. Πριν από ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκίνησε και προώθησε, έριξε αυτή την ιδέα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και υποθέτω ότι έγινε αυτό από πλευρά τη Ευρώπη, θέλω να πω, επειδή δεν πετύχαμε του στόχου τη Λισαβόνα και έπρεπε να βρεθεί ένα τρόπο για να καταφέρουμε να έχουμε υπό έλεγχο τους νέους στόχους, να τους θέσουμε υπό ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα το 2020 τελικά. Παρότι λοιπόν έχουμε στόχους και θέτουν τα κράτη-μέλη αυτούς τους στόχους από πλευρά τους, εκείνα τα ίδια είναι που ξεκινούν, αν μου επιτρέπετε, τις παραβάσεις ε, και παραβιάσεις. Ε. Και όπως είπε ο κύριος ε, ο συνάδελφος Τάκουλα, υπάρχουν αρχικές πρώιμες ενδείξεις από τα κράτη-μέλη για τους εθνικούς στόχους, για τις πέντε, τους πέντε τομείς που είχαν συμφωνηθεί υπό την στρατηγική για το 2020. Οι στόχοι για την εκπαίδευση και κατάρτιση, όλοι από αυτούς δεν έχουν προχωρήσει και έχουν υποβαθμιστεί και να δούμε σε σχέση με το 2020 οι στόχοι αυτοί δεν, δεν επαρκεί με αυτούς τους στόχους να σημειώσουμε μόνο αυτούς τους στόχους αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αποτυγχάνουν οι εθνικοί στόχοι στο να ανέθουν, να ανταποκριθούν σε αυτούς τους στόχους. Όπως και αποτυγχάνουμε στο να καταφέρουμε να έχουμε το αναγκαίο ποσοστό των πτυχιούχων μέχρι το 2020. Πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν περαιτέρω μέτρα και άμεση ρύθμιση και επανόρθωση από τα κράτη-μέλη. Ζητούμε να γίνουν αυτά από τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω μετά από ένα χρόνο σε ποιο επίπεδο θα βρίσκονται οι συζητήσεις μας. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα αποδώσει και υπάρχει αισιοδοξη πρόπτικη για τις δικές μας διεκδικήσεις. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, από ό,τι γνωρίζω από το βιο, βιωματικά από τις χώρες που πλήττονται υπάρχουν ε, μειώσεις ε, σε σχέση με τις ικανότητες από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βοηθήσει αυτό να πετύχουμε τους στόχους μας και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δικής μας Επιτροπής για την αντιστοίχηση των στόχων στην παιδεία και κατάρτιση. Είναι ένας πολύ σημαντικός ε, παράγοντας για τη διεύρυνση της καινοτομίας στην Ευρώπη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης που θα συνδέονται με τις νέες τεχνολογίε. Και πρέπει αυτό να το δούμε. Είχαμε και προ προηγούμενες συζητήσεις επ' αυτών. Δεν βλέπω όμως αυτή τη στιγμή πώς θα μπορέσει να υπάρξει αντιστοίχηση με τις σημερινές πολιτικές για την παιδεία και την κατάρτιση. Συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις ε, της ε, Προέδρου μας, κυρίας Πακ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτές τις παρατηρήσεις. Αν δούμε πραγματικά τους αριθμούς και τις δεσμεύσεις για την ε, παιδεία και κατάρτιση, την εκπαίδευση συνολικά, δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Σας ευχαριστώ. Thank uh, ευχαριστώ. Ναι, και εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πράγματι και ο πολιτισμός πρέπει να παίξει ένα πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Υπονομεύεται ο ρόλος του πολιτισμού από όλες τις μειώσεις πιστώσεων σε πάρα πολλές χώρες, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες οικονομικές. Στην δική μου χώρα πάρα πολλά προγράμματα απογυμνώθηκαν οικονομικά θα έλεγα και χρειάστηκε ορισμένα να σταματήσουν πλήρως. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε την κληρονομιά μας απέναντι σε αυτά τα προγράμματα λιτότητας. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι δυνατότητες χρηματοδότησης μπορούμε να έχουμε και από τον ιδιωτικό τομέα Βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα του πολιτισμού χώρες οι οποίες είναι σε δεσμευτικά προγράμματα συνεργασίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σαν παράδειγμα. Ευχαριστώ. Πρέπει να προσέξουμε να μην εντάξουμε όλα μας τα αιτήματα σε αυτό το κείμενο. Εδώ αυτό το κείμενο πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την, για την οικονομική πολιτική. Και δεν είναι δεν είμαι ευτυχής για όλα αυτά που σκεπτόμαστε και έχουμε ως φιλοδοξίες να τα εντάξουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλα υποχρεωτικά. Πρέπει να είμαστε κάπως πιο σύνετοι και αυτοπιθαρχημένοι. Δεν θεωρώ για παράδειγμα, Χάνο Τάκουλα, ότι το σημείο 7 όπως έχει μπορεί να παραμείνει έτσι με αυτή τη μορφή. Δεν πιστεύω ότι ένα πτυχίο πανεπιστημίου ποσοστό 40% πτυχιούχων πρέπει να πετύχουμε. Δεν υπάρχουν μόνο οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων που μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόλογο επίτευγμα. Αν βρίσκεται κάτι τέτοιο σε σχέση με την αυαρχίδα μας και το έχουμε αυτό, οι νέοι με, ένα, με, τα, και τα πανεπιστήμια ή παρόμοιες ισοδύναμες ε, δυνατότητες για τους νέους πάλι καταλήγουμε σε εκείνους που έχουν μια άλλη εναλλακτική δυνατότητα να τους θεωρούμε δεύτερης ποιότητας, δεύτερης κατηγορίας. Εκείνους που ασχολούνται με, τις, ε, ε, με την επαγγελματική κατάρτιση και γίνονται ειδικοί μάστορες σε κάποιο επάγγελμα και αποκτούν τον τίτλο του μάστορα και αυτοί λοιπόν δεν πρέπει να υποβαθμίζονται και να θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας επειδή δεν έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα. Κατά τα άλλα ευχαριστώ θερμά για τις παρεμβάσεις σας. Θα ήθελε η Επιτροπή να πει κάτι. Υπάρχει κάποιος, η κυρία Φιωρέλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε τον λόγο αν θέλετε παρακαλώ. Ε, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτά τα οποία γράφει Συμμεριζόμεθα εν πολύ στι απόψει τις οποίες εκφράζει, θα λάβουμε υπόψη το περιεχόμενό του. Θα ήθελα να υπογραμμίσω όμω ότι αν και είναι αλήθεια ότι η εκπαίδευση δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στι 10 κατά προτεραιότητα δράσεις τη ετήσια έκθεση, η ετήσια αυτή η έρευνα για την ανάπτυξη καλεί τα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε δαπάνες οι οποίες θα βοηθήσουν την ανάπτυξη στην εκπαίδευση ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα το 2011 και 2012 και ιδιαίτερα δύο προτεραιότητες υπογραμμίζονται, οι τέσσερα καθιστώντας την εργασία πιο ελκυστική και η πέντε επιστροφή των ανέργων σε θέσεις απασχόλησης. Και εκεί ε, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την προώθηση των επαγγελματικών ικανοτήτων. Και επίσης να μην ξεχνάτε και την προτεραιότητα 7 ε, ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια στην εργασία και στην ευελιξία και ελαστικότητα της εργασίας. Ε, για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να υπάρχει ε, ελεγχόμενη διαδικασία εκμάθησης και κατάρτισης των εργαζομένων ή των υποψηφίων εργαζομένων. Λοιπόν, έχουμε πάντα στο νου μας, νομίζω και με πλήρη τρόπο, την εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Ανωτάκουλα για τη δουλειά που έκανε. 14 Ιουνίου, καταληκτική προθεσμία, όχι 16 Ιουνίου. Εκπνέει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Τον Ιούλιο θα ψηφίσουμε προς έγκριση. Περνάμε τώρα σε συνάδελφο Κώστα. Προετοίμασε γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σίλβια, έχει τον λόγο, παρακαλώ. Η κυρία Σίλβια Κώστα, έχει τον λόγο. Ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσπάθησα στην έκθεσή μου να δείξω, να φέρω στην επιφάνεια την, τη σημασία που έχει η πλατφόρμα για την φτώχεια. Ο σύνδεσμος ε, του πολιτισμού από τη μία με τη μείωση της φτώχειας και την αντιμετώπιση της φτώχειας από την άλλη. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να επενδύσουν περισσότερο, να αναλάβουν περισσότερες υποχρεώσεις στον τομέα της παιδείας, της κατάρτισης και γενικά στην προσπάθεια ανύψωσης των επιπέδων εκπαίδευσης, όπως μας υπενθύμησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγαλύτερη προσπάθεια καταπολέμησης της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου ακόμα και από τα παιδιά που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα είναι ένας βασικός τρόπος για τη μείωση και της φτώχειας η οποία υπάρχει σήμερα και την βελτίωση της προσπάθειας αντιμετώπισης της. Να υπενθυμίσω εδώ την υποχρέωση που έχει αναλυθεί για την προσπάθεια σύγκρισης των διαφόρων πλαισίων τα οποία υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Εδώ υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση η οποία με τη σειρά της θα φέρει μια καθυστέρηση στην κινητικότητα των εργαζομένων. Ένα μια περαιτέρω πρόταση είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την αναπαραγωγή της φτώχειας από τη μία γενιά στην άλλη δίδοντας εγγυήσει ε, από την ε, ε, πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μέσω επίσης του αθλητισμού που θα επιτρέψει στα παιδιά να αποκτήσουν ικανότητες και νοοτροπίες οι οποίες θα τα βοηθήσουν στο μέλλον. Ένα άλλο θέμα είναι να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με διαπολιτισμικό τρόπο, στην εκπαίδευση εννοώ, για να βοηθήσουμε την ένταξη των παιδιών των μεταναστών στις χώρες μας, σε όλα τα επίπεδα της παιδείας. Θυμίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τον σημαντικό ρόλο που παίζει η εθελοντική εργασία, που μπορεί να βοηθά ε, τους νέους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν στη ζωή. Σχετικά με το θέμα της ένδυας νομίζω κάτι το οποίο έχουμε πει επανειλημμένα μέχρι τώρα και το έχει πει και η Πρόεδρός μας είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν τα λιγότερο ευνοημένα παιδιά σε οικονομικό κυρίως αλλά όχι μόνο επίπεδο στα πλαίσια του Youth on the Move σαν παράδειγμα. Να προσπαθήσουμε επίσης και διαγενειακές πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε την αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενιές, να καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα των γενεών και μέσω του συντονισμού των προσπαθειών των νέων. Θα ήθελα να προτείνω επίσης να προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε τις γνώσεις και τις ικανότητες φτωχών ανθρώπων, των φτωχών, γιατί δεν θα πρέπει να ταυτίζουμε ένα φτωχό πρόσωπο με κάποιον ο οποίος δεν έχει να προσφέρει στην κοινωνία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και οι φτωχοί και οι γυναίκες που βρίσκονται σε κακή οικονομική κατάσταση είναι σε θέση να προσφέρουν σε επίπεδο όχι μόνο φυσικά ικανοτήτων και αρμοδιοτήτων αλλά σε επίπεδο κοινωνικού πλούτου. Εν πάση περιπτώσει η αρχική έκθεση έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία εκφράζονται με πολύ σύντομο συνοπτικό τρόπο νομίζω ότι θα μπορέσουμε τελικά να καλύψουμε όποια και να υπάρχουν και να έχουμε πλέον τη βάση επί της οποίας ε, να ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας. Προβλέπεται σαν παράδειγμα και μια ενασχόληση με την εξωτερική διάσταση της καταπολέμησης της φτώχειας στα πλαίσια των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Εν πάση περιπτώσει τέτοια είναι τα θέματα τα οποία θα ήθελα να θέσω. Ελπίζω να σας ικανοποιεί η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σον Κέλλη. Εδώ μιλάμε για, την... για το πραγματικό νόημα της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ε, ειρήνη και την ευημερία όλων των πολιτών μας. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτά τα ζητήματα προκειμένου να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους ή ώστε των περισσότερους πολίτες. Και όταν ο κύριος ε, στόχος είναι να μειώσουμε τον αριθμό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Γιατί δυστυχώς πέφτουν μετά πολύ πιο εύκολα στην παγίδα της φτώχειας. Ε, αλλά και είναι πολύ πιο σε σε διάφορες κακές συνήθειες όπως ε, η χρήση ναρκωτικών ουσιών ε, ή η βία. Παρά την οικονομική ύφεση, οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να μειώσουν τις δαπάνες τους σε αυτό το τομέα. Είναι κέρια σημασία σε αυτό το θέμα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η βελτίωση των ε, ε, δεξιοτήτων, ε, των προσόντων των καθηγητών και των προτύπων ποιότητας, γιατί όσο καλύτεροι είναι οι καθηγητές τους, τόσο καλύτερα θα εκπαιδευτούν και αυτοί οι μαθητές. Πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που συμπεριέλαβε την πτυχή του αθλητισμού ως σημαντική πτυχή για την ε, ε, προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Δεν έχει αναγνωριστεί αρκετά αυτό κατά το παρελθόν και εδώ αναφέρεται στο σημείο 4. Ε, η εθελοντική εργασία αναφέρεται επίσης ως παράγοντας καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της, κοινωνική της κοινωνικής συνοχής και βεβαίως βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Θεμελιώδου σημασία λοιπόν όσα αναφέρονται. Και η πρόκληση εδώ για μας είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να, να εφαρμόσουμε και να ελοποιήσουμε τους στόχους που αναφέρονται στη στρατηγική για το 2020. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπίσκι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αξιοπρόσεκτη θα έλεγα. Αυτά που είπε η κυρία Κώστα μπορώ να τα προσυπογράψω όλα, αλλά έχω και μια σκέψη με όλα αυτά. Η κοινωνική φτώχεια δεν είναι πολιτισμική φτώχεια, ερώτηση. Θέλω να το θίξω αυτό, διότι είμαστε η Επιτροπή Πολιτισμού στην Ευρωβουλή. Εντάξει. Και η συνάντηση μεταξύ κοινωνικής φτώχειας και πολιτισμικής φτώχειας στις μικρές πόλεις μπορώ να το κατανοήσω, αλλά σε αυτόν τον κύκλο δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό, διότι έχουν όλοι αρκετά βιώματα και πείρα σε αυτόν τον τομέα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τίθεται για μένα το ερώτημα, Πρόεδρε. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, δεν είναι δυνατόν μέχρι αύριο να γίνει αυτό, ένα είδος πολιτισμικών ελάχιστων προδιαγραφών να απαιτήσουμε επειδή ακριβώς ε, έχουμε αυτή την προοπτική στρατηγική μέχρι το 2020 για τους νέους, ποιες ελάχιστες προδιαγραφές πρέπει να διασφαλιστούν σήμερα ώστε να μπορέσει κάποιο να διαφύγει από τη φτώχεια ή για του ενήλικες να μπορούν κάτι να, γίνει να κάνουν για την ανάπτυξη και προώθηση των παιδιών τους. Στα επιμέρους κράτη, αυτό συνδέεται αποκλειστικά τι πιο πολλέ φορέ με το ερώτημα πόσα χρήματα έχετε ή ποιοι θεσμοί υπάρχουν σε ένα χωριό ή σε μια πόλη. Διαδραματίζουν αυτά ένα ρόλο, αλλά δεν είναι ο μόνο και αποφασιστικό ρόλο. Θα το χαιρέτιζα ω Επιτροπή Πολιτισμού θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε πολιτισμικά ποιε είναι οι ελάχιστε προδιαγραφέ για του ανθρώπου και κυρίω για τα παιδιά στην Ευρώπη. Τι πρέπει να γίνει για να, είμαστε ανθρω... να δείξουμε ανθρωπιά και να είμαστε ανθρωπιστέ. Τι πρέπει να κάνουμε και πώ. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο, χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο, την αγαπητή συνάδελφο για τις ε, προτάσεις της. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φτώχεια είναι το υπαριθμόν ένα ε, σημείο που, από το οποίο θείται κανείς τον κοινωνικό αποκλεισμό και το βλέπουμε σε δύο σκέλη και στους Ευρωπαίους πολίτες και στους νεόπτωχους που έρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης. Επομένω, θεωρώ πολύ σημαντικό το άρθρο 5 για την ε, πρόθεση της ένταξης των μεταναστών και στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση. Δύο ερωτήσεις. Το σημείο 9, ε, τι εννοείται με τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, πώς εμπλέκονται δηλαδή στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων εκπαίδευσης οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και στο σημείο 10 θα ήθελα λιγάκι να μου διευκρινίσετε τη χρήση του όρου των φτωχών ανθρώπων. Ε, αναρωτιέμαι αν υπάρχει καμία, ένας άλλος όρος προκειμένου να περιγράψουμε ακριβώς αυτή την κατηγορία που ακούγεται λίγο στα ελληνικά τουλάχιστον, ακούγεται κάπως ε, ήδη κοινωνικά αποκλεισμένων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε έναν άλλον όρο. Δεν είμαι έτοιμη να σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Now, Hanno. Σε ευχαριστώ. Χάνο Τάκουλα παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Για την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ή ευρωπαϊκής δράσης που θα μπορούσαμε να συγκροτήσουμε. Και από πλευρά τη ε, ε, κυρία Ανέσκου, ω ε, σκιώδο εισηγήτρια και για όλου και για ω σκιώδη εισηγητή, θα ήθελα και εγώ να πω κάτι. Αυτό έχει οδηγήσει σε κάποιο προβληματισμό και κάποιες σκέψει από πλευράς συναδέλφου. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι υπήρξε έντονη ύφεση και σημειώνεται ισχυρή ύφεση στην Ευρώπη οικονομικά σε αυτή τη συγκυρία. Και ναι, ναι, ζούμε, βιώνουμε αυτή την ύφεση, όμως παρόλα αυτά, από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη ανήκει στις πιο πλούσιες περιφέρειες, περιοχές του κόσμου. Είναι και η πιο πλούσια κιόλα ίσως Ήπειρος. Και αν δει κανείς τα διαφορετικά στατιστικά στοιχεία, τι βλέπει από αυτά κανείς. Συμβαίνει λοιπόν ότι 18 εκατομμύρια βρίσκονται στο όριο, ζουν, βιώνουν το όριο της, στο της φτώχειας και βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλά παιδιά, απειρά παιδιά στο όριο της φτώχειας. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Αυτό οι νέοι, τα παιδιά, είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μιας κοινωνίας. Και όταν ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ε, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι για να κάνουμε κάτι. Και έχουμε το θέμα της παιδείας, της εκπαίδευσης που είναι το κλειδί για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Δεν επαρκεί, δεν επαρκεί το ποσοστό εκείνων που εγκαταλείπουν τα σχολεία πρόωρα να το καταφέρουμε να πιεστεί κάτω από τα 10%. Το θέμα είναι ποιος παραμένει τη μέση του δρόμου, στα μισά και δεν τα καταφέρνει. Πρέπει να βοηθήσουμε να μπορούν να ολοκληρώσουν και να προχωρήσουν οι νέοι. Είναι σημαντικό για μας να μπορεί στο πλήρες, στις πλήρες διαστάσεις να δημιουργηθεί αυτή η προσφορά. Δεν κάνω λόγο για μια κυδαιμονία που θα δημιουργήσουμε μια θέση κυδαιμόνα ή πατριού, πατριαρχικά να επιβάλλουμε κάτι. Όχι. Θέλουμε να προτρέψουμε, να ενθαρρύνουμε προς την παιδεία και εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να είναι δυνατόν από κοινού να ε, σχεδιάσουμε και να καταρτήσουμε μέτρα τα οποία θα σχεδιάσουμε και θα εγκριθούν. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να πω για το ποιος βρίσκεται σε μια σπυροειδή, καθοδική σπυροειδή εξέλιξη. Μπορεί κανείς να τα δει κανείς όλα αυτά. Το θέμα είναι αν έχει κάποιος τη βούληση να αντιδράσει και να λάβει μέτρα και να ενεργοποιηθεί. Υπάρχει η πολιτική βούληση νομίζω στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Σημαντικό είναι να μην την έχουμε μόνο αυτή την βούληση αλλά να περνάει προς το έξω το, προς το, το μήνυμά μας να κάνουμε κάτι ώστε τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν. Σας ευχαριστώ. Η Καταρίνα παρακαλώ έχει τον λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ και εγώ λέει η Καταρίνα. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που μόλις προανέφερε ο συνάδελφος, ότι το κλειδί είναι η παιδεία, η εκπαίδευση, το κλειδί για την επιτυχία. Είναι η μόνη πορεία, μονόδρομος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση ή δυνατότητα. Σημαντικό είναι να υποστηρίξουμε αναβαθμισμένο επίπεδο εκπαίδευσης και παιδείας. Η δυνατοτητα σημαντικο ειναι να υποστηριξουμε αναβαθμισμενο επιπεδο εκπαιδευσης και παιδειας η Πολύ καλά τα παρουσίασε στην πρότασή της όλα αυτά. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια επιπρόσθετα στοιχεία. Η φτώχεια πολύ συχνά έχει πρόσωπο γυναικείο. Πολλές φορές είναι τα νέα κορίτσια εκείνα που δεν έχουν επαρκή προσόντα, δεν έχουν επαρκώς εκπαιδευτεί και δεν έχουν τα αναγκαία προσόντα και καταλήγουν έτσι στο να παραστρατήσουν ή χάνουν τον ίσιο δρόμο. Ας το πω έτσι. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι δραστηριότητες, εξωσχολικές δραστηριότητες, πάρα πολλές φορές βασίζονται σε εθελούσια βάση, εθελοντικά και για τα θέματα για μια κοινωνική ένταξη των παιδιών στις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τέτοιου είδους δραστηριότητες πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά και στους νέους, ώστε να έχουν το αίσθημα ότι είναι εισάξιοι και ισότιμοι πολίτες με, με τους άλλους. Θα πρέπει η ψηφιοποίηση του διαδικτύου το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει προαχθεί σημαντικά ακριβώς μέσω του διαδικτύου υπάρχουν πολύ καλές δυνατότητες τα παιδιά, οι νέοι να προχωρήσουν στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση, να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις δράσεις. Αυτά που ανέφερε πιο πριν ο κύριος Μπίσκι. Πώς μπορεί κανείς με τον πολιτισμό να καταπολεμήσει τη φτώχεια. Σημαντικό στοιχείο. Το Υπουργείο Παιδείας σε εμά στη χώρα μας δίνει για τέτοια παιδιά ας το πω έτσι, κουπόνια. Κουπόνια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες πολιτιστικές ε, εκδηλώσεις. Για να πηγαίνουν στο θέατρο, σε θεατρικές παραστάσεις, στον κινηματογράφο με αυτά τα κουπόνια τα παιδιά. Και να μην ε, χρειάζεται, επειδή οι γονείς τους δεν έχουν τα χρήματα να στερηθούν αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και να μπορούν να τις παρακολουθήσουν έτσι. Ευχαριστώ. Yeah. Ε. ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να πει κάτι. Έχω εδώ ποιος είναι, ο κύριος Χάντους, παρίσταται ή όχι. Δεν χρειάζεται να παρέμβει, λέει. Εντάξει. Η κυρία Κώστα θα ήθελε να πει δύο λόγια. Παρακαλώ Σίλβια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, διάφορες ε, προτάσεις που εκφράσατε εδώ. Ε, με τα χαρά ε, να εμπλουτίσω την γνωμοδότηση αυτή με τις προτάσεις σας. Η γνωμοδότηση θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική εν ώψη ε, δεδομένου μάλλον το ότι η στρατηγική για το 2020 δεν εστιάζει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε στις, ε, στους κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού. Καλό είναι λοιπόν να το πράξουμε τουλάχιστον τώρα. Σε ό,τι φορά το άλλο σχόλιο του κυρίου Κέλλη, βεβαίω και το είχα ε, συμπεριλάβει σύντομα, αλλά σε μια περίοδο κρίσης, όπως είπε και ο κύριος Στάκουλα, υπάρχουν δεσμεύσεις ε, μεταξύ των οποίων και στη δική μου χώρα, ε, που ενδεχομένως να μας οδηγήσουν σε περικοπές ε, στις ε, δαπάνες για, την, για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, αυτό που ανέφερε ο κύριος Σοβίσκη για τα ελάχιστα πολιτιστικά κριτήρια, ελάχιστε πολιτιστικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές, είναι δύσκολο να τις ορίσουμε. Μπορούμε όμως να ορίσουμε τις βασικές δεξιότητες, μεταξύ των οποίων οι δεξιότητες των πολιτών. Ε, υπάρχει και έκθεση για αυτό το θέμα. Ε, μπορούν να υπάρχουν υπάρχουν δεσμεύσει, μάλιστα ε, από όλα τα κρατημέλη για να δημιουργήσουν συγκεκριμένε ενδείξει. Ε, κύριε Παλιαδέλη, για τι ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει, πολλέ χώρε έχουν την εξή εμπειρία. Όχι ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει μπορούν να υποκαταστήσουν το Υπουργείο, αλλά ότι μπορούν να το ενισχύσουν, να συμπληρώσουν το έργο του με την εμπειρία του ε, στη δεύτερη ευκαιρία, σε αυτό το σύστημα τη δεύτερη ευκαιρία. Ε, πολλοί άνθρωποι κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σύστημα, να αποκτήσουν νέε δεξιότητε και νέα προσόντα. Επίση, οι οργανώσει ε, των νέων με εθελοντές πολλές φορές διδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην, ε, στην ενθάρρυνση των ε, παιδιών ε, σε ό,τι αφορά, την παροχή κινήτρων σε ό,τι αφορά το σχολείο. Τώρα, για τον όρο φτωχός. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε έναν, έναν όρο μεταξύ μας για να κατανοούμαστε. Εγώ μίλησα για φτώχεια και έτσι μετά έκανα λόγο και για φτωχούς. Όμως, ουσιαστικά μιλάω για την περιθωριοποίηση. Πολύ ε, συχνά υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ ε, της απώλειας ε, δεξιοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού ή της περιθωριοποίησης. Ο κύριος Τάκουλα ανέφερε αυτό το τραγικό αριθμητικό στοιχείο. 20 εκατομμύρια παιδιά κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Επίσης αναφέρθηκε ε, στο ενδεχόμενο ε, μετάδοση της φτώχειας από γενιά σε γενιά. Ε, πρέπει να αξιοποιήσουμε βέβαια στο σχολείο και την οικογένεια που είναι και τον πολιτισμό μάλλον που είναι οχήματα για την κοινωνική πρόοδο και άνοδο. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στο σχολείο σε όλα τα παιδιά, ακόμα και τα παιδιά με αναπηρία. Συμφωνώ απολύτως λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμη μια τροπολογία επ' αυτού του ζητήματος προκειμένου να δεσμευθούν τα κράτη-μέλη να θέσουν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους ε, για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της ε, ε, εγκατάλειψης του σχολείου. Η Κατρίνα μίλησε για την ε, για το γεγονός ότι όλο και περισσότερο γυναίκες ε, ε, ζουν κάτω από το έργο της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Και θα πρέπει βεβαίως να σκεφτούμε και την διαβίου μάθηση και την εξαποστάσεως μάθηση προκειμένου να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να επιστρέψει στο χώρο της εκπαίδευσης έχουμε να κάνουμε και με επίπεδα φτώχεια τα οποία δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς, άειλης εν πολύ φτώχεια. Και γι' αυτό θα πρέπει να ανοίξουμε όλες τις πόρτες της ενσωμάτωσης της κοινωνικής και της κατάρτισης και των ε, διδασκόντων βέβαια που παίζουν σημαντικό ρόλο για να μπορέσουν να επαναφέρουν σε σωστό δρόμο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σας ευχαριστώ πολύ Καταρίνα. Σίλβια θέλω να πω, όχι Καταρίνα, συγγνώμη. Όπως είπαμε, τον Ιούνιο θα έχουμε καταληκτική προθεσμία στις 14 Ιουνίου κατάθεση τροπολογιών. Τον Ιούλιο θα ψηφίσουμε για να εγκρίνουμε. Και περνάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης τώρα. Ανταλλαγή απόψεων με την Culture Action Europe. Η κυρία Κίση είναι παρούσα, η οποία μπορεί άμεσα να παρουσιάσει την εισήγησή της. Δεν θα χάσουμε χρόνο. Παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ξεκινήστε. Πείτε μας τι κάνετε ως Culture Action Europe. Τι κάνετε σε σχέση με τα θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς. Παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ κυρία Πακ. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής σας. Αντιπροσωπεύω το Culture Action Europe, μια πλατφόρμα που εκπροσωπεί πολλές ΜΚΟ για τον πολιτισμό στην Ευρώπη σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιους τρόπους υποστηρίζεται ο πολιτισμός στην Ευρώπη σήμερα. Η εκστρατεία ονομάζεται «Είμαστε παραπάνω, είμαστε περισσότερο». θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην σημαντική συνεισφορά την οποία προσφέρει ο πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση γενικότερα. Τώρα ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχουμε, δεν θα, δεν θα εκπλαγείτε. Έχουμε δύο βασικούς στόχους. Ο ένας είναι ένα τολμηρό πολιτιστικό πρόγραμμα και δεύτερο να υποστηρίξουμε με τον πιο σημαντικό δυνατό τρόπο τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με δημοσιονομικά. Αλλά προσπαθούμε εμείς να επηρεάσουμε και τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές πλαίσιο και θα θέλαμε οι νομοδοτήσεις της Επιτροπής σας να γίνονται δεκτές. Αναφερόμαστε σε αρκετές ε, εκθέσεις και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Μπαρόσο. Απαιτείται βέβαια να έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία να μπορέσει να μας βοηθήσει να λειτουργήσουμε με πιο φιλόδοξο τρόπο. Από την βδομάδα αυτή έχουμε μαζέψει 10.000 υπογραφές και πιστεύουμε να φτάσουμε τις 20.000 μέχρι το μήνα Ιούλιο. Αυτές τις υπογραφές θα σας τις καταθέσουμε και σαν απάντηση στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό και για τη συνάντηση των Υπουργών Πολιτισμού που θα ακολουθήσει το φθινόπωρο. Η δική σας δουλειά εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος. Θέλουμε να βοηθήσουμε στις προσπάθειές σας, αλλά γενικότερα ελπίζουμε ότι και τα μέλη της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου θα, θα υπογράψουν συγγνώμη, το συγκεκριμένο μανιφέστο και έτσι θα μπορέσετε κι εσείς να καταλάβετε τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε και ελπίζουμε η υπόθεση του πολιτισμού να μην χαθεί στους επόμενους γύρους διαπραγμάτευσης για τα δημοσιονομικά. Στην έρευνα της Eurostat για το 2009 είδατε ότι το 90% του πληθυσμού της Ευρώπης πιστεύει ότι οι ανταλλαγές οι πολιτιστικές είναι πάρα πολύ σημαντικές και γι' αυτό στον τομέα αυτό θα θέλαμε να συλλέξουμε τις ιδέες σας έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και την επόμενη χρονιά. Συνεπώς λοιπόν, αν συνδυάζουμε τις προσπάθειές μας, θα αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι παραπάνω από μια οικονομική ένωση. Ελπίζω η παρουσίασή μου να ήταν ενημερωτική και συνοπτική βέβαια. Ήθελα να επενθυμίσω μόνο ότι η οργάνωση που αποκαλείται σήμερα European Forum, Ευρωπαϊκό Φόρουμ. Όχι, Culture Action Europe ονομάζεται σήμερα αυτή η οργάνωση. Τη γνωρίσαμε ήδη το 1992 υπό το τίτλο European Forum for Arts and Heritage, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνών και κληρο... Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και έτσι συνεργαστήκαμε πολύ στενά από τότε. Υπενθυμίζω την τελευταία φορά, στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία, είχαμε αυτή την εκστρατεία για τα κέντρα για πολιτισμού και δεν ε, έφταναν τα χρήματα και οι εκδηλώσει ούτε από τη μία ούτε από την άλλη κατεύθυνση. Μπορώ να σας διασφαλίσω για το γεγονός ότι σας ε, έχει αποσταλεί ένα βίντεο σε σχέση με τον Παρόζο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά στο Σώμα των Επιτρόπων μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα έχουμε την οροφή των δημοσιονομικών προοπτικών και με αυτή πρέπει σε αυτή να προσαρμοζόμαστε. Γνωρίζετε όμως πάντα ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπαμε ότι υπάρχουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υποστήριζαν και υποστηρίζουν το έργο μας. Έχουμε περιορισμούς. Οι περιορισμοί μας είναι τα κονδύλια που μας δίνουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω, αλλά προσπαθούμε στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων να θέσουμε νέα κέντρα βάρους και βασιζόμαστε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως σύμμαχο όταν θα αναλαμβάνει, θα έχει αναλάβει το αξίωμά του και όχι ως ιδιώτη, ως πολίτη, να μας δοθούν περισσότερα κονδύλια στο μέλλον. Διότι αποκτήσαμε το βίωμα, την πείρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο πολιτισμός είναι και αυτός ένας συντελεστής οικονομικός, οικονομικός παράγοντας. Με αυτά τα επιχειρήματα μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ περισσότερους για τα θέματα πολιτισμού. Και είναι καλό να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πέρα από το ότι είναι ωραίο είναι καλό λοιπόν. Έχουμε όμως περιορισμούς, δεν μπορούμε όλα να τα κάνουμε. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να εγγραφούν και να υποστηρίξουν τα άτομα που είναι υπέρ ημών και μπορούν να είναι σύμμαχοί μας και να συνεργαστούν μαζί μας πρέπει να τύχουν της υποστήριξή μας και να τους την προσφέρουμε. μου δημιούργησε κάποια μηχανία η σύγχυση το σύνθημά σας, διότι έχει συχνά αναφερθεί, υπάρχει ο κύριος καθηγητής Εβερντινγκ, Γερμανός που απεβίωσε δυστυχώς πριν από 15 χρόνια σε μια διάσκεψη είχε πει στο ερώτημα τι είναι πολιτισμός απάντησε ο πολιτισμός είναι το παραπάνω αυτό το οποίο είναι ένα συν το επιπλέον. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Είναι το ίδιο σε σχέση με το δικό σας σύνθημα. Το ίδιο νόημα έχει. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να λάβει τον λόγο. Υποθέτω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα έλεγα απόψε θα καταλήξουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, θα προσυπογράψουν και θα δώσουν υποστήριξη με αυτόν τον τρόπο στο έγγραφο αυτό, στην πρωτοβουλία αυτή. Εντάξει, και αν κάποιο δεν μπορεί να το κάνει, οι συνεργάτες να ζητηθεί να το κάνουν εκείνοι για λογαριασμό τους, ώστε να μπορέσει να προαχθεί αυτό, να γίνει αυτό. Και οι δικοί μου εξασκούμενοι σταζιέρ το κάνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία και Είναι μια εξαιρετική ιδέα. Είναι κάποιο από την Επιτροπή εδώ. Η κυρία Μαγνούν, όχι, δεν παρίσταται. Θα ήθελα να τη πω, ο κύριο Μπαρόζο υποσχέθηκε κάτι το οποίο δεν μπορεί να τηρήσει, ε. Τέλο πάντων, εντάξει, έστω. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά, Κυριακή. Είμαστε στο πλευρό σα, σύμμαχοι. Και για τα επόμενα προγράμματα θα μεριμνήσουμε για όλα αυτά. Κλείνει αυτή η σημαντική συνεδρίαση τώρα. Περνάμε στη συνάντηση συντονιστών τώρα. Όλοι που δεν είναι συντονιστέ μπορούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα και να πάνε σε άλλη, απασχόλη, σε άλλη ασχολία του. Ευχαριστώ. Τέρμα η συνεδρίαση λίγη. Ευχαριστώ.